έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα, παράλληλα με την προστασία των ζώων. Και γι' αυτό, ως εισηγήτρια, θέλω να σας προτείνω να απορρίψουμε αυτές τις τροπολογίες που προτείνονται. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ψηφοφορία. Αν γίνουν αποδεκτές αυτές οι τροπολογίες, η θέση μας δεν θα είναι ε, σωστή. Όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, ε, σίγουρα αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να ξανανοίξει αυτό το θέμα, δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε τις ίδιες ε, εργασίες, δεν θα εξυπηρετούσε ούτε την προστασία των ζώων κάτι τέτοιο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που θα ήταν θετικό είναι το να κλείσουμε αυτό το φάκελο τώρα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι ε, που μπορούν να το επιβεβαιώσουν και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και σήμερα να χειριστούμε σωστά αυτό το θέμα και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι θετικό για την προστασία των ζώων και για την έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Grazie, Ευχαριστώ πολύ, Ελίζαβετ. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία, θα δώσω τον λόγο στον Λουίς Καμπλασάντος. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η έκθεση αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί μας δημιουργεί σοβαλά συνειδησιακά προβλήματα. τα δικαιώματα των ζώων είναι πολύ παρόμοια με τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι δύσκολο να συμφιλιώσουμε την επιστημονική χρήση των ζώων και την αποφυγή αγωνίας και ε, πρόκληση αγωνίας και πόνου σε αυτά τα, τα πλάσματα. Νομίζω ότι ο συμβιβασμός όμως είναι καλός, είναι ο εφικτός ε, ε συμβιβασμός και εμείς θα τον υπερψηφίσουμε, θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Νομίζουμε ότι ο συμβασμός, επαναλαμβάνω, είναι θετικός, δεν χρειάζεται να ξανανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ, Λουίς. Εάν ε, δεν υπάρχουν άλλοι... Α, ναι, η κυρία Πάλουσεν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Γέγκλε. Πρόκειται για την ε, καλύτερη δυνατή ε, συμφωνία την οποία επιτύχαμε. Θέλαμε να συμφιλιώσουμε την προστασία των ζώων αφενός ε, και την επιστημονική έρευνα αφετέρου. Οι φιλελεύθεροι λοιπόν θα ψηφίσουν κατά την έννοια των ενδείξεων της συγγετρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πόλσεν. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι. Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα στην ψηφοφορία. Έχετε μπροστά σας τον κατάλογο των τροπολογιών. Διανατάσεως της χειρός. Όχι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γι' αυτό λοιπόν ψηφίζουμε τώρα για την τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχέ Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Ο Αλμπέρτο πήγε να κάνει λάθος. Αποχές απορρίπτεται. Τέλος, τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Αποχές και η τροπολογία 5 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τελική ψήφος επί των συστάσεων της δεύτερης ανάγνωσης υπέρ. Κατά. Καμία ψήφος κατά. Αποχές τέσσερις αποχές. Και επομένως μπορώ να πω ότι, ε, Ελίζαμπετ, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ε, με την εργασία αυτή, γιατί και, και εσύ πρέπει να είσαι ικανοποιημένη. Η εργασία σου έγινε αποδεκτή από την πολύ μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αλλάξουμε λίγο, θα αντιστρέψουμε λίγο την ημερήσια διάταξη. Ακούστε με λίγο. Μία μικρή αντιστροφή λοιπόν, γιατί ο κύριος Βοτζιεβόσκι, ο αντιπρόεδρός μας, θα φύγει σε λίγο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε τώρα με το σημείο 8, ε, βάσει του οποίου θα πρέπει ο συνάδελφος Τσόφσκι να μας ενημερώσει σχετικά με την επίσκεψη της επιτροπή Επιτροπής μας στην Ρουμανία. Θα του δώσουμε λοιπόν αμέσως τον λόγο. Φτάσαμε στο σημείο 8 ε, έτσι ώστε να προλάβουμε να μας κάνει την ενημέρωση ο κύριος Βοζγεχόφσκι. Ευχαριστώ. 12 μέλη της Επιτροπής μας επισκέφθηκαν τη Ρουμανία πριν από δύο εβδομάδες. Η επίσκεψη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε την Γεωργία στη Ρουμανία από κοντά. Η Ρουμανία είναι καινούριο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο μέλος από το 2007 και μετά. Και ήταν πράγματι πολύ χρήσιμη ευκαιρία να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Ίσως δεν είναι μια χαρακτηριστική χώρα σε ό,τι αφορά το γεωργικό τομέα, γιατί η πλειοψηφία του αγροτικού, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο το είδαμε από κοντά. Νομίζω ότι η κατάσταση στη Ρουμανία είναι αντιπροσωπευτική της κατάστασης των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, φίλους από τη Ρουμανία, την κυρία Τανσίλα, την κυρία Σάρμπου, που οργάνωσαν, διοργάνωσαν τα, περισσότερε από τι εκδηλώσει τις οποίε παρευρεθήκαμε κατά τη διάρκεια τη επισκέψή μα, Η οργάνωση ήταν εξαιρετική και μας δόθηκε η ευκαιρία σε τρεις μόνο μέρε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Η πιο σημαντική εκδήλωση ήταν η συνάντηση με το στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Συναντηθήκαμε με Ρουμάνους πολιτικούς υπεύθυνου για τη Γεωργία. Με τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Ντουμήτρου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, της Ρουμα... Ρουμανικής Γεωργίας επίσης, καθώς επίσης και με εκπροσώπους των Ρουμανικών Συλλόγων και Ενώσεων Γεωργών της Ρουμανίας, εκπροσώπων του γεωργικού τομέα εκπροσώπους των γεωργικών επιχειρήσεων, των ίδιων των γεωργών, των αγροτών κλπ. Η ερμανική γεωργία περνάει δύσκολες στιγμές. Προσπαθεί απλώς να, να επιβιώσει, όχι να αναπτυχθεί. Πολεμάει για την επιβίωσή της. Αγωνίζεται να ζήσει. Οι συνάδελφοί μας στη Ρουμανία μας είπαν ότι περίπου το 1 τρίτο της γης δεν καλλιεργείται αυτή τη στιγμή και το διαπιστώσαμε η διεισόμαση. Το 1 τρίτο της γης είναι εγκαταλελειμμένη και αυτό είναι χαρακτηριστικό στα νέα κράτη-μέλη. οι άμεσες πληρωμές είναι πολύ χαμηλές και γι' αυτό το λόγο η γη εγκαταλείπεται και η κατάσταση στην πλησία των εκμεταλλεύσεων είναι πολύ δύσκολη. Είδαμε ε, μια εκμετάλλευση 50 εκτάριων με 15 αγελάδες και 70 πρόβατα. με την Ελίζαμπεθ επισκεφθήκαμε μαζί αυτήν την εκμετάλλευση και στρέφουμε και προς ε, εκείνη γιατί πράγματι ε, η εντύπωση που προέκυψε ήταν ότι αποτελεί σημαντικό, σημαντική πρόκληση για μας και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο ε, τις μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. εκμεταλλεύσεις όπου ολόκληρη οικογένεια εργάζεται εκεί. Και ταυτόχρονα προφυλάσσει και προστατεύει το περιβάλλον. Η επίσκεψη ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Είναι ένας ε, τύπος γεωργίας αυτή η οικογενειακή ε, γεωργία σε μικρές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να υποστηριχτεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια... Α, όχι, έχουμε την Ελίζαμπετ. Μπέτ. ganz... Κυρία Γέγκλε, Ήθελα προς, προς την κυρία Τανσίλα και τους δύο συναδέλφους να τις ευχαριστήσω θερμά γιατί μας προετοιμάσταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα ήταν ότι ε, το 1 τρίτο της επιφάνειας, της γεωργικής επιφάνειας ε, δεν καλλιεργείται ε, και αυτές οι επιφάνειες, αυτές οι εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται. Είδαμε στην επίσκεψή μας ότι ήταν στην Τρανσιλβανία σε κάποιες περιοχές που υστερούν σε σημεία όπου υπάρχουν μικροί γεωργοί και που θα έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να καλλιεργούνται. Σε αυτά τα σημεία στα οποία κάναμε την επίσκεψή μας φάνηκε ότι ε, οι αγρότες και οι οικογένειές τους ε, ταλαιπωρούνταν και προσπαθούσαν ε, να τα βγάλουν πέρα όσο μπορούσαν. Και γι' αυτό μου δημιουργήθηκε το ερώτημα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και παράλληλα να αποφύγουμε το, να μην χορηγούνται ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μόνο σε μεγάλες επιφάνειες Πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο για την άσκηση της γεωργικής πολιτικής. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, για μένα, να δούμε τη διάκριση μεταξύ του αγώνα του μικρού καλλιεργητή και των μεγάλων επιφανειών. Molto bene, grazie. Άψογα, ευχαριστούμε Ελίζαμπετ. Ποιος άλλος, κάποιο άλλος έχει δει στο λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με αυτό το θέμα το οποίο πολύ σωστά αναφέρθηκε και ήταν και το κύριο έβριμα της αντιπροσωπείας. Χρήση γης και άμεσες πληρωμές. Θα ήθελα να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν κάποιες τροπολογίες ε, σχετικά με το μέλλον της ε, ΚΑΠ μετά από το 2013. Υπήρξε μια σημαντική τροπολογία η οποία λέει για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις άλλες ε, πιο νέες χώρες ε, θα εξισωθούν ε, οι άμεσες ε, πληρωμές intended before 2006. θα εξισωθούν λέω μέχρι το 2016 idea is the, the direct payment. στο 100%. Ε, και ε, επομένως ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε οτιδήποτε άλλο και να κινηθούμε στην ίδια γραμμή. Το 2013 είναι μεθαύριο, θα πρέπει τα κριτήρια να είναι ίδια, είναι καλά κριτήρια και για τους γεωργούς και για τους ε, καταναλωτέ. Βεβαίω καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε του καταναλωτέ, αλλά καταλαβαίνετε ότι κάποια νέα κριτήρια θα είναι πολύ δύσκολα για του γεωργού και μικρότερες πληρωμές με περισσότερα και με υψηλότερα κριτήρια, αυτό θα δυσκολεύσει πάρα πολύ τους ε, γεωργούς και επομένως ε, πιστεύουμε ότι πριν από το 2016, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να φτάσουν οι άμεσες πληρωμές στο 100%. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Και τώρα, εάν δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις ε, σχετικά με την παρουσίαση του Γιάννου Βοτσεβόσκη, να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως, Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο. Οι διεθνείς συμφωνίες ε, για το εμπόριο, και ζητώ την προσοχή σε συνάδελφοι, ε, καθώς επίσης και η απελευθέρωση των ανταλλαγών στην Γεωργία έχουν σοβαρό αντίκτυπο στους ε, γεωργούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Οι σχέσεις με τον ΠΟΕ, ε, συμπεριλαμβανομένων και των διαπραγματεύσεων της ΕΝΤΟΧΑ έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε άμεσα μηχανισμούς αντιστάθμισης για τους παραγωγούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης, Επίσης ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, οι επιπτώσεις ε, των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανταγωνιστικότητα, σε την προστασία γενικότερα και του πρωτογενούς τομέα αλλά και του διατροφικού τομέα, αλλά φυσικά και άλλα στοιχεία όπως είναι η ευζοία των ζώων, η αηφόρος ανάπτυξη, η προστασία προϊόντων ποιότητας κτλ. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλία με εισηγητή τον κύριο Παπαστάμκο. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, θεωρήθηκε μια, ε, μια ε, επίσης συνδεδεμένη επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 50 του κανονισμού και έχει οριστεί σχετικό έγγραφο καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Επιτροπών Άγκρη και Ίντα. Η Επιτροπή Ανάπτυξη, καθώ επίση και η Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντο, τη Δημόσια Υγεία και τη Ασφάλεια των Τροφίμων, ορίστηκαν ε, για εκπόνηση γνωμοδότηση. Κύριε Παπαστάμκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προσυπο... Προσυπογράφω τα όσα αναφέρατε εισαγωγικά ε, ασχοληθήκαμε και επιψηφίσαμε την έκθεση Lion για το μέλλον της κοινή αγροτικής μετά το 2013 αλλά όπως πολύ σωστά σημειώσατε η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει και την, τις εξωτερικές της πτυχές, έχει την εξωτερικότητά της η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, επηρεάζεται αν θέλετε από παγκόσμια ή διμερή ή διαπεριφερειακά ρυθμιστικά καθεστώτα και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση είναι η άλλη πλευρά, το αναγκαίο συμπλήρωμα της ε, έκθεσης ε, Λάιον για την ε, εσωτερικότητα της κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 2013. Λίγα στοιχεία στην αρχή που καταδεικνύουν ακριβώς τη σημασία του, της έκθεσης με τίτλο Διεθνές, Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο, Ευρωπαϊκή Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο. Το Παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών αγαθών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ του 2000 και του 2009. Γνώρισε δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης, 25% το 2007 και το 2008. Βεβαίως το 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης, έγιναν εμφανείς οι επιπτώσεις και στο εμπόριο γεωργικών αγαθών. Είχαμε μία μείωση 3% κατ' όγκων και 13% καταξίαν. Ε, πρόκειται για επιπτώσεις οι οποίες ήταν οι ποιότερες σε σχέση ε, με άλλους κλάδους. Ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των γεωργικών αγαθών. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σημείωσε ιστορικό χαμηλό το 2005, 27 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισε εμπορικό πλεόνασμα 4,5 δισεκατομμύριων ευρώ, επανήλθε όμως το στο ελληματικό, σε ελληματικό εμπορικό ισοζύγιο το 2007 2,4 δις Το 2008 άγγιξε επίπεδα ρεκόρ ε, καθώς το έλλειμμα ανήλθε σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009 μειώθηκε ξανά σε 2,5 δις ευρώ, γεγονός που οφείλεται στο ότι η οικονομική κρίση έπληξε λιγότερο τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε για μείον 8% σε αξία και περισσότερο τις εισαγωγές, μείον 13%. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριαρχούνται από τελικά προϊόντα, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 2 τρίτα, 68% της αξίας των εξαγωγών ε, και αναφέρουμε στο διάστημα 2007-2009, με τον Ίνο το κρασί να βρίσκεται στην πρώτη θέση οι 12 από τις 15 κατηγορίες σημαντικότερων εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν τελικά προϊόντα. Τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα εμπορεύματα, τα commodities, αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως 23% και 9% των εξαγωγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε εξαγωγικό μερίδιο αγοράς το 2008 από το 19% το 2007 βρέθηκε στο 18% το 2008. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών αγαθών με το μερίδιο επί των παγκοσμίων εισαγωγών να ανέρχεται περίπου στο 20%. Τα πέντε κυριότερα προϊόντα που εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το άλευρο σόγιας, ο καφές, η σόγια, οι μπανάνες και το κακάο με τις περισσότερες εισαγωγές να προέρχονται από μερικούς βασικούς προμηθευτές. Υπογραμμίζεται ότι το άλευρο σόγιας και η σόγια αντιπροσωπεύουν το 12% των συνολικών εισαγωγών με προμηθευτές στη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις ΗΠΑ. Το εμπόριο πρωτογενών και μεταποιημένων γεωργικών αγαθών αντιστοιχεί περίπου στο 6% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Το μερίδιο το 1995 ήταν 9%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη δυναμική αύξηση 150% στο εμπόριο βιομηχανικών αγαθών κατά τα τελευταία έτη. Όσον αφορά τις αγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, η και μας διασυνδέει την ε, προσέγγιση την οποία κάνω με την παγκόσμια εμπορική κλίμακα και ιδίω με τις διαπραγματεύσει του γύρου της Δόχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων, παραλαμβάνω από τις αναπτυσσόμενες χώρες, η αξία των εισαγωμένων αγαθών ανήλθε σε 83 δισεκατομμύρια δολάρια στο διάστημα 2007-2009, είναι περίπου το 70% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο, περισσότερες εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από, από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία από κοινού στις άλλες προηγμένες βιομηχανικά χώρες. Στην έκθεση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρουν στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Αντικείμενο εξέτασης θα είναι αφενός οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ και η γεωργική προσφορά, το, offer, το γεωργικό offer της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γύρο της Δόχα και αφετέρου οι διμερείς διαπεριφερειακές εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης με τρίτες χώρες. Ε, θέλω να πω την προσωπική μου άποψη και να πιστεύω ότι συμμερίζονται και άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα αυτή ότι είναι ιδιαίτερος ανησυχητική η στάση της Κομισιόν και αναφέρομαι στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Εμπορίου στο ντοσχέ του Διεθνούς Εμπορίου και όχι στην, ε, στο ντοσχέ της Γεωργίας και στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση ως προς τις γεωργικές παραχωρήσεις στις οποίες προβαίνει. Στο πλαίσιο η Κομισιόν προέβη πολύ νωρίς, ε, Οκτώβριος του 2005, σε πολύ εκτεταμένη προσφορά, σε πολύ εκτεταμένο offer στο γεωργικό τομέα, προκειμένου να αποσπάσει από τους εμπορικούς σετέρους εταίρους παραχωρήσεις στους τομείς των βιομηχανικών προϊόντων, ΝΑΜΑ και των υπηρεσιών. Είχα ζήσει από κοντά όλη αυτή την ε, γενναιόδορη στάση της ε, Κομισιόν γιατί ήμουνα και στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι διαπραγματεύσει του γύρου τη Δόχα στο Χονγκ Κονγκ. Θα εξετάσουμε επίση την έκθεση τι διμερεί διαπεριφερειακέ συμφωνίε, όπω και τι ολοκληρωθήσει διαπραγματεύσει των συμφωνιών που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ. Αναφέρομαι στι συμφωνίε με το Μαρόκο, την Νότιο Κορέα, το Περού και την Κολοβία, τι χώρε τη Κεντρική Αμερική. Κατά τη γνώμη μου, οι συμφωνίε που διαπραγματεύτηκε η Κομισιόν και οι γεωργικές παραχωρήσεις στις οποίες προέβη έναντι τόσο των χωρών των Άνδεων όσο και έναντι των χωρών της Κεντρικής Αμερικής δημιουργούν εύλογες ανησυχίες. Μεταξύ άλλων, ενδεικτικά αναφέρω τις αδεσμολόγητες ποσοστώσεις στους τομείς της ζάχαρης και του ρυζιού. Οι λόγω ποσοστώσεις ξεπερνούν τις παραγωγικές δυνατότητες των χωρών αυτών με εμφανή τον κίνδυνο της ανάπτυξης τριγωνικού εμπορίου απούσεις, δηλαδή την ώρα που απουσιάζει, μία ρήτρα καθαρού εξαγωγέα. Παράλληλα θα εξετάσουμε και τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις και αναφέρομαι προφανώς τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μερκοσούρ και τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και δύο σε ορισμένους τομείς. Υπογραμμίζω μεταξύ άλλων το ήδη άκρος ελληματικό εμπορικό ισοζύγιος βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων καθώς και την ελληπή συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, παραδείγματο χάρη στον τομέα του βοήου κρέατος. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην άκρος, συνδετέρως άκρος περιοριστική πολιτική που ασκεί η Αργεντινή ως προσαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες, παρακολύοντας την έκδοση πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας. Τα μέτρα αυτά έχουν ήδη πλήξει τις εξαγωγές πολλών ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων. Και επιτρέψτε να πω ότι απίφθηνα ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Επίτροπο Ντεγούχτ στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Αν δηλαδή η Κομισιόν έθεσε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων που ε, ε, έγινε πριν από 15 μέρες στο Buenos Aires ε, στην πρώτη φάση όπως είπα των διαπραγματεύσεων και αν αυτό το θέμα εγείρει ζητήματα ασυμβατότητας των μέτρων της Αργεντινής με τους κανόνες και τις πειθαρχίε του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της Κομισιόν και την απουσία διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και ιδίω ως προς τις γεωργικές πτυχές. Θα εξετάσουμε ακόμη τα προβλήματα που ανακύπτουν ως προς την αποτελεσματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης από τρίτες χώρες. Ειδικότερα θα αναλυθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Παγκοσμίου ε, Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και οι πρόνοιες, οι προβλέψεις σε διμερείς συμφωνίες. Στις ολοκληρωθήσεις διαπραγματεύσεις λόγω χάρη με τις χώρες των Άδεων και της Κεντρικής Αμερικής, το παράρτημα των προστατευόμενων γεωργικών ενδείξεων περιλαμβάνει πολύ μικρό αριθμό των συνολικών ΠΟΠ και ΠΓΕ ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την παγκόσμια θεσμοθετημένη εμπορική μεγακλίμακα, πέραν των κανόνων του ΠΟΕ και του γύρου της Δόχα, θα μελετήσουμε και τις επιπτώσεις που έχουν επιφέρει στον ευρωπαϊκό γεωρικό τομέα αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων, των πάνελς του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Εμπορίου. Λόγω χάρη, και θυμίζω ε, την, ε, τη, τη, μεταρρύθμιση, τη ριζική μεταρρύθμιση της ΚΟΑ Ζάχαρης που έγινε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θετία, ότι είχε ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση από καθαρό εξαγωγέας να μετατραπεί σε καθαρό εισαγωγέα ζάχαρης. Επίσης, λόγω της απόφασης στην υπόθεση σχετικά με το ορμονούχο βόηο κρέας, ήταν τεράστιων αντιμέτρων στις ευρωπαϊκές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Στον στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ως γνωστόν, εκκρεμεί ακόμη, κατόπιν αμερικανικού αιτήματο, η υπόθεση σχετικά με τα χλωριωμένα πουλιαρικά και αυτό θέτει ζήτημα προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών, ζήτημα θέμη του ανταγωνισμού στους εχώριους παραγούς, εάν επιτρέπαμε την εισαγωγή χλωριωμένων πολυερικών. Ξεχωριστή σημασία έχει τέλος το ζήτημα των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας και της αποτελεσματικής εισαγωγής των εισαγωμένων προϊόντων σε ισοδύναμους, σε αντίστοιχους κανόνες. Είναι πρωτίστως ζήτημα προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αλλά είναι συγχρόνως και ζήτημα προστασίας των παραγωγών μας, των Ευρωπαίων παραγωγών, από τον αθέμετο ανταγωνισμό που υφίστανται λόγω της αθρώας εισαγωγής προϊόντων που υπάγονται σε πολύ ελαστικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτά ως μια πρώτη προσέγγιση, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, του ε, θέματος που μας αποσχολεί, της ε, Έκθεση την οποία καλούμαστε, ε, καλούμε να επεξεργαστώ. Προσβλέπω στη συνεργασία όλων των πτερίγων της Επιτροπής μας και προκειμένου, και το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια, να αναδείξουμε κοινού τόπους όπως αρμόζει σε μια Επιτροπή η οποία ασχολείται, έχει στο επίκεντρό της, του λειτουργικού πεδίου αρμοδιότητά της, την ε, ε, Ευρώπη της, της και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εμάς κύριε Πρόεδρε, όσο και τους συντονιστές όλων των ομάδων, ιδιαίτερα τον κύριο Ντες, για την τιμή που μου κάνετε να μου αναθέσετε αυτό το πολύ σημαντικό, πολύ ευαίσθητο ε, φάκελο, ε, ο οποίος τυκλοφορείται ε, ε, γεωργία και διεθνές εμπόριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαστάμικο. Βεβαίω συμφωνούμε μαζί σου, η Ευρώπη έγινε πλέον μια περιοχή του κόσμου ε, με πολύ μεγάλο αριθμό και όγκο εισαγωγών γεωργικών προϊόντων όσον αφορά τις τριγωνικές πωλήσει και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να απασχολήσει οπωσδήποτε την ε, Επιτροπή μας. Όσον αφορά τώρα την ονομασία προέλευσης, προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης και επ' αυτών θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Πολλοί έχουν εγγραφεί για να πάρουν το λόγο. Η κυρία Μαγκίνης, παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίαση που μας έκανε. Λίγα σχόλια. Κάναμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο μια συζήτηση για το θέμα τη Μερκοσούρ. Μη ικανοποιητική συζήτηση όσον αφορά τη δική μα επιτροπή. Έγινε μια κοινή συζήτηση. Δεν μου είχε ζητηθεί η γνώμη μου εκ των προτέρων για να πω αν συμφωνούσα ή όχι. Και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου και με την διοργάνωση και με τις απαντήσεις που λάβαμε, γιατί νομίζω ότι δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες του γεωργικού τομέα και αυτό θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά, ότι η Επιτροπή δεν απάντησε στις ερωτήσεις που θέσαμε εμείς. Μια δεύτερη παρατήρηση για το πώς εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας ε, μπαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Φαίνεται ότι έχει προτεραιότητα η Επιτροπή Εμπορίου και μετά το ανακαλύπτουμε εμείς και τότε αρχίζουμε να μπαίνουμε στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εξεταστεί, γιατί υπάρχει μια κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη, υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα για τις περιοχές της Υπέστρου και θα πρέπει οι δικές μας ανησυχίες να αντικατοπτρίζονται σε εμπορικές συμφωνίες, είτε του ΠΟΕ, είτε διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Νομίζω ότι η κατάσταση σε σχέση με την Αργεντινή και το αν μπορούν να αρχίζουν και να σταματούν τις εμπορικές ροές όποτε θέλουν είναι επικίνδυνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν έχουμε συμφωνίες με τέτοιου είδους χώρες, επικίνδυνη για θέματα διατροφικής ασφάλειας ε, και άλλα. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Θα εξετάσω την έκθεση αυτή προσεκτικά και θέλουμε η έκθεση αυτή να εκφράζει τις ανησυχίες που έχουμε για τη γεωργία. Και το θέμα των προτύπων και των ετοιμάτων μας είναι κάτι που πρέπει να συζητείτε σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, σε εμπορικές συμφωνίες. Προς το παρόν δεν είναι αντικείμενο αυτών των εμπορικών συμφωνιών και αυτό πρέπει να αλλάξει διότι η αγρότες στην Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνίζονται με εισαγωγές τρίτων χωρών όταν έχουν υψηλότερα στοιχεία κόστους από ό,τι για την παραγωγή σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ και θα περιμένουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Λουίς Κάπουλας Σάντος έχει ζητήσει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαστάμκο για τα λόγια του. Εκ μέρους της ε, σοσιαλιστικής ομάδας ε, θέλω να δηλώσω ότι είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί του για ένα θέμα τόσο σημαντικό για μας. Είδα τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2010 και διαπιστώνω ότι ε, παρόλο που ε, έχει μειωθεί η συνολική αγορά κατά 2,2%. Ε, υπάρχουν όμως χώρες όπως η Ινδονησία, η Κορέα που έχουν αυξήσει τις εξαγωγές κατά 7,5%, αντίστοιχα η Βραζιλία 4,5%, ε, η Κίνα 2,7% κλπ. Ε, παρόλο λοιπόν ότι υπάρχει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες ε, αυξάνουν τις εισαγωγές τους, συγγνώμη, τις εισαγωγές τους και θα, μπορούσε, θα μπορούσαν να είναι σημαντικοί πελάτες μας ε, και να απορροφήσουν δικές μας εξαγωγές. Ε, από την άλλη μεριά θα πρέπει να αποφύγουμε εμείς να γίνουμε οι συνδικαλιστές του τομέα, αλλά θα πρέπει να γίνει μια υπεύθυνη και έξυπνη συζήτηση για να προασπίσουμε τα συμφέροντα της γεωργίας μας χωρίς να πληγούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση λαϊκισμού, ε, βολονταρι, βολονταριστική συζήτηση που τελικά θα οδηγήσει στο να πλήξουμε αυτό που το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε. Είναι λοιπόν πολύ ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερο ενδιαφέροντο το θέμα αυτό και πολύ ευαίσθητο. Ευχαριστώ πολύ, Λουίση. κύριε Λαβία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παπαστάμκο για αυτήν την ε, εισαγωγή που έκανε στο θέμα, αλλά και γιατί μας έδωσε μια, μια σειρά στοιχείων που θα μας δώσουν την δυνατότητα να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό και να προωθήσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να διευρύνω λίγο τις σκέψεις που έκανε αναφερόμενος σε στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα ε, ε, εισαγόμενα προϊόντα. Γιατί η ιστορική πραγματικότητα καταδεικνύει ότι παραδοσιακά η Ευρώπη είναι εισαγωγός προϊόντων ε, κατά κανόνα, κακάο, καφέ και άλλα προϊόντα διατροφής τα οποία δεν παρήγονται στην Ευρώπη. Όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία διευρύνουν τα προϊόντα. Και επομένως αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεγάλες εισαγωγές προϊόντων που όμως παράγονται και στην Ήπειρό μας. Και επομένως εδώ υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού και άρα το ζήτημα είναι πιο ευαίσθητο και θα πρέπει οπωσδήποτε με κοινοτικές ε, αποφάσεις, με αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπιστεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, νέα συγκεκριμένα μέτρα και εξηγώ γιατί. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός υφίσταται πολλαπλές πιέσεις και σίγουρα από πιέσει θα δούμε πολλέ όταν θα, μιλά, θα ε, συζητήσουμε για την κοινή γεωργική πολιτική. Και επομένω μπορούμε με ευκολία να εισάγουμε αντισταθμιστικά μέτρα έτσι ώστε να αντισταθμιστούν κατά κάποιο τρόπο οι ζημίε των γεωργών αυτών που θα ζημιωθούν ιδιαιτέρω από διμερεί ή πολυμερει συμφωνίε. Θα ξεκινήσει λοιπόν μία ε, ένας αγώνας ε, που ε, στην ουσία όμως θα παραμείνει λίγο στα χαρτιά. Ήδη μπορώ να φανταστώ από τώρα τις συζητήσεις στην Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, για αντισταθμιστικά μέτρα όσον αφορά τις μπανάνες ας πούμε. Για τρίτη τέταρτη φορά συνεδριάζουμε για να μιλήσουμε για την απελευθέρωση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού. Όμως τελικά δεν φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Ε, αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία να εξευρεθούν συμπληρωματικοί πόροι. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη περιθωρίου δράσης και αντίδρασης. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν αυτό το πλαίσιο, ε, χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένες και δυνατές προτάσεις. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν ε, να ξεχάσουμε την ανταγωνιστικότητα των δικών μας γεωργών. Θα πρέπει η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών μας ε, να παραμείνει σταθερή. Δεν είναι δυνατόν να τους πιέζουμε διαρκώς και να υφίστανται εκείνοι διαρκώς τις ε, κακές ε, επιπτώσεις, ε, τις αρνητικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού. Θα πρέπει βεβαίως όλοι όσοι εισάγουν προϊόντα στην Ευρώπη να σέβονται τους κανόνες που σέβονται ήδη οι δικοί μας γεωργοί. Όσον αφορά επίσης την σωστή αντιμετώπιση της παραγωγής, όσον αφορά τις σωστές συνθήκες, όσον αφορά τους ηθικούς κανόνες, τους κανόνες δεοντολογίας, είναι είναι πολύ συγκεκριμένα ε, τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να εισάγουμε προϊόντα που αποτελούν ε, αποτέλεσμα εργασίας ε, μικρών παιδιών. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δεχτούμε εισαγωγές προϊόντων που δεν έχουν παραχθεί με σεβασμό των ορθών κανόνων. Ευχαριστούμε πολύ, Εσ, και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο, τον κύριο Παπαστάμκο, για την έκθεση που μας παρουσίασε και για την παρουσίαση της κατάστασης στον τομέα του εμπορίου και της γεωργίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να εξαγάγουμε. Είναι σαφές ότι δεν θέλουμε προστατευτισμό, θέλουμε ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερο εμπόριο με κανόνες το απόλυτα ελεύθερο εμπόριο δεν λειτουργεί. Πολλές φορές έχουμε δώσει το εξαιρετικό παράδειγμα των χρηματοοικονομικών αγορών με τις τεράστιες ζημίες που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι για τη διασφάλιση της αγροτικής οικονομίας και του γεωργικού μοντέλου στην Ευρώπη να φροντίσουμε σε διμερείς, σε πολυμερείς συζητήσεις ε, στον ΠΟΕ να προάγουμε και να διασφαλίσουμε αυτό το γεωργικό μας μοντέλο. Και η κυρία Μακίνες ε, ε, είπε ότι δεν ήταν ικανοποιημένη με τις απαντήσεις της Επιτροπής. Και εγώ, Μέιριντ, δεν ήμουν ικανοποιημένος από τις απαντήσεις, αλλά δεν ήμουν ικανοποιημένος ούτε από τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Και άκουσα από το περιβάλλον του Επιτρόπου ότι ε, και ο Επίτροπος ε, εξεπλάγει σχετικά με ε, τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα που έχουμε πάρει και από την Λισαβόνα και να δούμε ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα γεωργικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στη βιωσιμότητα ενώ σε πολλές ε, περιοχές ε, ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε βιώσιμη ε, γεωργία και εκτίθενται πολλές περιοχές στο εμπόριο χωρίς να είναι βιώσιμη, βιώσιμο το γεωργικό μοντέλο. Θα πρέπει με τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτουμε να λάβουμε υπόψη μας τους κινδύνους που υπάρχουν. Έχουμε ανοίξει τα σύνορά μας για πολλές ε, χώρες του κόσμου και υπάρχουν πολλές οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ε, θρησκευτικέ οργανώσεις που φροντίζουν για τις τρίτες χώρες και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν γιατί δεν υπάρχουν ίδιες συνθήκε σήμερα όπως πριν από 20-30 ε, χρόνια. Τα περισσότερα προϊόντα μας τα εισάγουμε από τον χώρο του τρίτου κόσμου, όπω είπε ο συνάδελφο κ. Παπαστάμκος, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των εισαγωγών μας. 90% των ε, προϊόντων ε, από την Αφρική. Ε, είμαστε εισαγωγή των 95% των προϊόντων, 44% των προϊόντων από την ε, Λατινική Αμερική. Είμαστε εισαγωγή προϊόντων από Αυστραλία, από Καναδά, από πολλές χώρες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το τι πολιτική θα ακολουθήσουμε. Εδώ Έχουμε σε αυτό το τομέα πολύ καλά επιχειρήματα και θα πρέπει να φροντίσουμε τη διασφάλιση της ποιότητας. Και στο Κοινοβούλιο πολλοί συνάδελφοι θα συμφωνήσουν επ' αυτού και δεν μπορούμε στην Ευρώπη να επιτρέψουμε κινδύνους για την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική μέσα από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. δεν θέλουμε ε, να προωθήσουμε το απόλυτα ελεύθερο μοντέλο, πρέπει να προωθήσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα παρέχει και κάποιες διασφαλίσεις. Και από εξαγωγής καφέ και μπανάνας ε, έχουμε παραδείγματα από 2,75 που ήταν η τιμή για τα 18 κιλά μπανάνες προσθέθηκαν 25 cents ε, ως επιβάρυνση και στο Ρότενταμ τελικά κατέληξε να κοστίζει 7 ευρώ και στα στα γερμανικά σούπερ μάρκετ ε, τελικά κατέληξε να πουληθεί αυτή η βαλίτσα 35 ευρώ. Αν δεν έχουμε δική μας παραγωγή στην Ευρώπη, διατρέχουμε τον κίνδυνο του πολύ υψηλού κόστους από εισαγόμενα ε, προϊόντα. Αυτό το έχουμε δει ε, με προϊόντα όπως η ζάχαρη και από χώρες όπως η Βραζιλία που θέλουν να κυριαρχήσουν στην ε, παραγωγή ζάχαρης παγκοσμίω. Χρειαζόμαστε διατάξεις που θα διασφαλίζουν το εμπόριο προς όφελος των καταναλωτών στην Ευρώπη, όχι μόνο προς όφελος της γεωργίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Στεφάν Λεφόλ, παρακαλώ. Σύμφωνο με τους προλαλήσαντες, τον κ. Σαντόσα, την κυρία και τον ε, Αλμπέρ, τον Αλμπέρτ. Νομίζω το τι μπορούμε να κάνουμε, το τι θα κάνουμε θα εξαρτηθεί από το πόσο μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, να κινητοποιηθούμε. Η Κομισιόν εδώ και 15 χρόνια χρησιμοποιεί διαπραγματευτικές ε, εντολές ε, με στόχο να ανοίξουμε ε, τη δική μας αγορά τη, γεωργικών προϊόντων, προκειμένου οι άλλοι να ανοίξουν τη δική τους αγορά για τα βιομηχανικά προϊόντα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Είμαστε ικανοί ε, στην εμπορική μας στρατική να εντάξουμε τη γεωργία. Και όταν ε, λέω γεωργία, μιλώ τα μεταποιημένα προϊόντα, τα αγροτροφημικά προϊόντα. Εμείς έχουμε τις δικές μας, είχαμε τις ε, δικές μας ευθύνες, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί όταν εξάγαμε με επιστροφές. Αυτό το σύστημα θα τελειώσει το 2013. Δεν μπορούμε όμως να κουβαλάμε αυτή την ευθύνη ε, στο μέλλον. Ε, να θεωρούμε ότι είμαστε ένοχοι πλέον. Εμείς στην Ευρώπη άλλωστε χρειαζόμαστε ένα αριθμό προϊόντων που θα τα παράγουμε εδώ. Το βόλιο κρέα, για παράδειγμα. Ήδη στην Γαλλία Κάποιοι το λένε. Δυσκολευόμαστε να βρούμε βόλιο κρέας στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Αρκετό ώστε να ικανοποιήσουμε την εσωτερική μας ζήτηση. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν τίθενται και η ικανότητά μας να βαρύνουμε έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η εντολή, δηλαδή υπέρ των υπηρεσιών, υπέρ της και εις βάρος της γεωργίας, η ικανότητά μας αυτή είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικό να εξασφαλιστεί. Γιατί οι βιομηχανοί και, και οι πάροχοι υπηρεσιών πιέζουν πάρα πολύ και θα πρέπει εμείς να αντισταθούμε όλοι μαζί. Και αν κάποια στιγμή ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει των ΠΟΕ, θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένω. Ε, ε, σε σχέση με το, τις διμερείς διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα, αλλά οι, οι διαπραγματεύσει των ΠΟΗ θα πρέπει να γίνουν με διαφορετική εντολή, όχι με την ίδια εντολή που ε, γινόντουσαν οι προηγούμενες τα 15 χρόνια. Γιατί στα υπερπόντια διαμερίσματά μας αυτή τη ε, στιγμή καταργείται ε, σιγά σιγά η παραγωγή της μπανάνας. Ε, τι θα παράγουν. Τους δίνουμε αντιστάθμιση, τους δίνουμε βοήθεια, αλλά αρκεί αυτό. Θα πρέπει κάτι να παράγουν κιόλα. Αυτή τη στιγμή πάγουν να παράγουν και μπανάνες. Κάτι πρέπει να παράγουν. Συνεπώ, συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ στιβαροί, να δώσουμε καθαρό μήνυμα προ την Κομισιόν, έτσι ώστε ο αγροτροφημικός τρομέας, η γεωργία, να ενταχθεί στην εμπορική μας πολιτική με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, όπου ανοίγαμε τη δική μας ε, αγορά γεωργικών προϊόντων προκειμένου να πάρουμε αντισταθμίσματα στην βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών. Θα πρέπει να κάνουμε το λογαριασμό κάποια στιγμή. Αυτό που χάσαμε στη γεωργία όλα αυτά τα χρόνια το κερδίσαμε στην βιομηχανία και στι ε, υπηρεσίε. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξουμε τη στρατηγική μα και αυτή θα ήταν η καλύτερη στρατηγική. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Μάρτιν και μετά στον Τζέιμ Νίκολσον. Ναι, νομίζω ότι σε πολλά σημεία συμφωνούμε και ευχαριστούμε τον κύριο Παπαστάμκο για την παρουσίαση που μας έκανε. Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα που έχουμε από διάφορες διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής που δεν είναι πάντοτε διαφανή και μπορεί να, φοβά, φοβόμαστε το ίδιο, ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις χώρες του Μερκοσούρ. Και οι απαντήσει τη επιτροπή δεν ήταν ικανοποιητικέ. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει η Επιτροπή τα προβλήματα που έχει η Γεωργία σε αυτό τον τομέα και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Το ελεύθερο εμπόριο σε επιχείρημα το είδαμε και από το χρηματοπιστωτικό τομέα, οπότε δεν χρειάζονται περισσότερα επιχειρήματα. Ποιο είναι ο στόχο που έχουμε για το εμπόριο, μα ενδιαφέρει ο ισολογισμό και οι εισαγωγέ. Αν δούμε τις εισαγωγές λεκυθίνης παραδείγματος χάρη, πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος παραγωγής στις χώρες της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη. Και στις εισαγωγές ε, πρέπει να τηρούνται όχι μόνο εμπορικά πρότυπα, αλλά και κοινωνικά ε, και οικονομικά ε, μοντέλα. Και τα πρέπει να συνεισφέρουν ε, στην ε, ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά. Ε, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να δίνουμε δισεκατομμύρια για το σύστημα, αλλά αν αφήνουμε τόσα πολλά ανοιχτά παραθυράκια, αν δεν διασφαλίσουμε εμεί τον οίκο μα, αν δεν διασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, αυτό θα είναι ει βάρο του ευρωπαίου παραγωγού, αλλά θα είναι ει βάρο και των παραγωγών στον τρίτο κόσμο τελικά. Πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μα. θα πρέπει σε ορισμένα σημεία να δείξουμε συνέπεια και όσον αφορά τι εξαγωγικέ επιστροφέ και η πολιτική μα ομάδα πολύ συχνά το έχει αναφέρει αυτό. Οι εξαγωγικέ επιστροφέ είναι κάτι το οποίο έχει σημασία για τη δική μα αξιοπιστία στο διεθνέ εμπόριο και οι πρακτικέ ε, τι οποίες εφαρμόζουμε νομίζω έχουν σημασία για τη δική μα αξιοπιστία και γι' αυτό το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να λήξουν οι πρακτικές που δεν μας ωφελούν. Ευχαριστώ. Thank you very much, President. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την συζήτηση τη περασμένης εβδομάδα είναι ευκαιρία να σκεφτούμε τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ε, περιμένω να συνεργαστώ με τον εισηγητή τους, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Ε, η απάντηση όμως του, σκόπου, του Επιτρόπου την περασμένη εβδομάδα ε, με ανατρίχιασε. Διότι είπε τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Εμείς στην Ευρώπη ορίζουμε κάποια πρότυπα, κάποιες προδιαγραφές με βάση τις οποίες η παραγωγοί, οι μεταποιητές και οι καταναλωτές ε, συμφωνούν. Τώρα, ο Επίτροπος τι λέει. Και είμαστε η Επιτροπή Γεωργίας, έτσι. Αντιπροσωπεύουμε την αγροτική βιομηχανία, τον αγροτικό τομέα. Μας είπε όμως, δεν με νοιάζει αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Εγώ θα προβώ στις συμφωνίες που θεωρώ κατάλληλες. Θα θα εισάγουμε ε, τροφές και ζώα στο, στην Ευρώπη ε, που δεν θα συμμορφώνονται με τα δικά μας πρότυπα και τις δικές μας προδιάφεσες. Αυτό μας το πολύ καθαρά. Νομίζω ότι έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόκληση. Ε, νομίζω ήταν πολύ υπεροπτικός ο, ο Επίτροπος όταν μας μίλησε και μας προκάλεσε, διότι εμείς τουλάχιστον έχουμε εκλεγεί ενώ αυτός δεν έχει εκλεγεί ό,τι και αν πιστεύει για μας. Λοιπόν, η Επιτροπή μας θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Να έρθει σε σύγκρουση μαζί του, διότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλές προδιαγραφές για τα τρόφιμα τα οποία θα εισάγονται στην Ευρώπη. Οι ίδιες με τις δικές μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δύο διαφορετικές προδιαγραφές, δύο διαφορετικά πρότυπα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά οτιδήποτε εισάγεται ω τρόφιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τι δικέ μα προδιαγραφέ. Αυτό θα πρέπει να το καταστήσουμε σαφέ στον Επίτροπο. Νομίζω δεν το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στα παρασκήνια, ε, τι ζημιώσεις ε, ε, γίνονται για να μας συρθούμε σε αυτή την συμφωνία με τη Μερκοσούρ, αλλά θα το καταλάβουμε στο μέλλον γιατί συνήθως ο, ο χρόνος ε, φωτίζει τις κρυφές ταυτότητες όλων. Θα το δούμε, θα περιμένουμε, θα το δούμε. Αλλά εμείς από την άλλη μεριά, εντωμεταξύ, θα πρέπει να ασκήσουμε το δικό μας δικαίωμα να προβάλλουμε και να προασπίσουμε τη δική μας άποψη. Όχι μόνο στο Μερκοσούρ, στη σχέση με το Μερκοσούρ, αλλά και στον ΠΟΕ. Διότι έχουμε ρόλο σοβαρό να παίξουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παπαστάμκο για την παρουσίασή του. Ε, σε γενικέ γραμμέ ε, συμφωνούμε με την άποψή του. Πρώτον, υπάρχει μια μεγάλη άγνοια για το ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στι διαπραγματεύσει του ΠΟΕ. Υπάρχει μια άγνοια από πλευρά κοινή νόμη και των καθημερινών ανθρώπων, των καταναλωτών. Οι καταναλωτέ αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν τι καταναλώνουν στις αγορές. Δεν έχουν ιδέα ούτε και καταλαβαίνουν ποιο θα είναι ο αντίκτυπος των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που ζητάμε από του Ευρωπαίου παραγωγού και δεν το ζητάμε από του παραγωγού άλλων χωρών. Συνεπώ θα πρέπει να φωτιστεί η πραγματικότητα. Ε, να γίνει γνωστή η κατάσταση. Ε, θα, το έγγραφό μας θα πρέπει να βοηθήσει τις οργανώσεις των καταναλωτών και γενικότερα την κοινή γνώμη να καταλάβει καλύτερα την κατάσταση. Ε, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ μακριά. Στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου πολύ συχνά συνάδελφοί μας αγνοούν τον αντίκτυπο των δικών τους αποφάσεων πάνω στη γεωργία. Ε, ίσως και εμείς θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα την άποψή μας ενδεχομένως. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί σήμερα να λέει, να μας πει ποια, είναι, ποια θα είναι η θέση της στον ΠΟΕ, αν θα βελτιώσει την προσφορά της ε, ε, ή αν θα ε, καταφέρει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και των ε, παραγωγών μας, τότε ε, θα μπορούσαμε και εμείς να προσθέσουμε μία ε, θέση, μία παράγραφο στην έκθεσή μας που θα προασπίζει τη θέση των παραγωγών μας. Χρειαζόμαστε αξιοπρέπεια και μία παραγωγή σε ίσους όρους με αυτή την παραγωγή των άλλων χωρών. Παραγωγή η οποία θα έρθει τελικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν με αυτά που θα στέλνουν και θα εξάγουν σε άλλες χώρες. Μας ενδιαφέρει αυτά που θα εξάγουν σε εμάς. Χρειάζεται να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, θα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τον πλανήτη όμως, όχι μόνο την, ε, τη, δική μας γωνιά εδώ στην Ευρώπη. Γιατί τι λογική έχει αν εμείς απαγορεύουμε φυτογενομικές ουσίες ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές να χρησιμοποιούνται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού ή στην Βόρεια Αφρική. Ε, αν είναι κακές για την υγεία θα πρέπει να είναι κακές για την υγεία όλων, όχι μόνο τη δική μας Λοιπόν, ε, αν είναι να χρησιμοποιούνται κατουσίε, α τι χρησιμοποιούν και οι δικοί μα. Δεν έχει νόημα να τι χρησιμοποιούν μόνο οι άλλοι Γεώργοι. Επίση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη δική μα άποψη στην, για την έκθεση ποιότητας, στην έκθεση για την ποιότητα ε, που ζητούσαμε να γίνει επισήμανση των προϊόντων για την προέλευση των συστατικών τους. Αυτό που θέλουμε ε, είναι απλώς, για παράδειγμα, να γραφτεί αν το προϊόν θα είναι, είναι κοινοτική προέλευση ή μη κοινοτική προέλευση. Αυτό αρκεί. Α δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε για ορισμένα απλά πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι διμερεί συμφωνίε με τρίτε χώρε. Αν δεν καταφέρνουμε να ελέγξουμε τη συμμόρφωση με τις ε, διμερείς ε, συμφωνίε, γιατί τι υπογράφουμε τι διμερεί συμφωνίε. Γιατί να υπογράψουμε μια καινούργια συμφωνία με το Μαρόκο, αν ποτέ δεν έχει κάνει σεβαστή μία, ούτε μία από τι ποσοστώσει των παλαιότερων συμφωνιών. Γιατί αφού δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τι παλιότερε συμφωνίε, να υπογράφουμε καινούργιε. Σε ό,τι δεν αφορά τι διαπραγματεύσει με τι χώρε τη Λατινική Αμερική, σίγουρα χρειαζόμαστε αυτέ τι αγορέ. Αλλά θα πρέπει να απαιτούμε ένα ελάχιστο ποιότητα προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των, των εργατικών εργασιακών δικαιωμάτων κλπ. Δεν είναι δυνατόν εμείς να ε, ξεπουλάμε τη δουλειά των δικών μα γεωργών επειδή αυτό το χρειάζονται μεγάλε μα εταιρείε σε άλλου τομεί. Ε, οι συμφωνίε αυτές πρέπει να δούμε αν μας δίνουν κάποιο κέρδο, κάποιο αποτέλεσμα. Ποτέ δεν έχουμε κάνει ένα απολογισμό. Και δεν μιλάω για τη Λιτανική Αμερική, με την Κίνα, α πούμε. Έχουμε κάνει ποτέ απολογισμό των συμφωνιών που έχουμε υπογράψει με την Κίνα. Έχουμε κάποιο όφελο από αυτέ ή όχι. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Μάτο και Δεν ε, παρόλο που είμαστε πρωταθλητέ κόσμου, δεν μου δίνετε το λόγο πιο νωρί. Τι αξίζει λοιπόν να είμαστε πρωταθλητέ κόσμου, δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων. Ε, θέλω να συγχαρώ, να συγχαρώ όσου είχαν την ε, πρωτοβουλία, ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή. γιατί θα χρησιμεύσει. θα χρησιμεύσει να εκφράσουμε τι ανησυχίε μα και να προβάλλουμε έναν τομέα που είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη. Ο κ. Παπαστάμικος έδωσε πολλά νούμερα, μίλησε για τη φιλοσοφία και μίλησε και για πολλά πράγματα τα οποία έχουμε, για τα οποία έχουμε επανειλημμένω μιλήσει σε αυτή την εδώ την Επιτροπή. Για τι ε, ε, συμφωνίες, ε, διμερείς και άλλε Πρέπει να δούμε τι συμφωνίε του ΠΟΕ, ε, ποιο θα είναι το εύρο του, Οι διμερεί συμφωνίε, για παράδειγμα, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Την έλλειψη διαφάνειας για την έλλειψη πληροφόρησης και είναι ένας πολύ άσχημος κοινός παρανομαστής. Ε, είμαστε υπέρ του γεωργικού μας τομέα, υπέρ της γεωργίας μας και της κτηνοτροφίας μας και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ασυμβίβαστο με την υποστήριξη των άλλων τομέων της οικονομίας μας και του διεθνούς εμπορίου. Παρόλο που ορισμένοι το παρουσιάζουν έτσι. Αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με αυτές τις εκθέσεις είναι το εξή. Σε σχέση με τον ΠΟΕ έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ποιο θα είναι το εύρος των διαπραγματεύσεων αν αυτές ξαναξεκινήσουν και τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στο μέλλον. Υπάρχει κάτι που με ανησυχεί ή σε σχέση με τις ε, ε, διμερείς συμφωνίες όμως. Γίνονται διαπραγματεύσεις και ε, δεν τις παρακολουθούμε. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα τους πριν το δούμε. Κολομβία και Περού για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, καλλιέργεια μιας, μια καλλιέργεια μόνο, η μπανάνα, να πληρώσει το τίμημα μια ολόκληρης συμφωνίας, τη οποία συμφωνίας δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τα ωφέλη εκ των προτέλων. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γάλλο συνάδελφο, για τους παραγωγούς μπανάνας. Και εμεί έχουμε παραγωγού στα Κανάρια. Α του αφήσουμε να παράγουν. Το κάνουν καλά και αυτό ξέρουν να κάνουν. Παράγουν τι πιο ποιοτικέ μπανάνε του κόσμου. Και ε, δεν θα ζητούσαν αντιστάθμιση, δεν θα ζητούσαν καμία βοήθεια αν οι συμφωνίε οι οποίε είχαμε καταλήξει με χώρε τη Λατινική Αμερική και άλλε δεν ήταν τόσο αρνητικέ. Λοιπόν, ναι, συμφωνίε, ναι, αλλά με ποιου όρου και του όρου να του ξέρουμε εκ των προτέρων. Αν οι όροι είναι καλοί, δεν θα χρειάζονται αντισταθμίσει μετά. Μετά, Μερκοσούρ. Ξεμπλοκαρίστηκε ε, η συμφωνία, η, η ανταπόκριση την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ήταν πολύ αρνητική, αυτό είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή ε, όμως τουλάχιστον γνωρίζουμε πριν την υπογραφή τη συμφωνία ποιο ήταν ο αντίκτυπο. Αυτό είναι σημαντικό. Για το Μαρόκο, να επαναλάβω ότι με το Μαρόκο δεν έχει νόημα να διαπραγματευτούμε καινούργια συμφωνία όταν δεν τηρείται η παλιότερη εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών. Ευχαριστώ. Grazie. Grazie. Ευχαριστώ πολύ. Μισελ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα στον εισηγητή για την παρουσίαση που μας έκανε. Και εγώ στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα γιατί ε, στα λόγια του ε, Επιτρόπου αισθάνθηκα μια κάποια αλαζονία. Ναι, αλαζονία. Γιατί δεν μπορεί να είναι άγνοια η αμάθεια ε, εκ μέρους του, άγνοια των γεωργικών θεμάτων. Βλέπουμε τα αριθμητικά στοιχεία, βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις της ανάπτυξης ε, στην Κίνα ή ε, σε άλλες χώρες και δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι η γεωργία θα αποτελέσει τον μοναδικό τρόπο συναλλαγής και αντισταθμίσματος στις συμφωνίες με τις χώρες αυτές οι αντισταθμίσεις δικαιολογούνται όταν υπάρχει ε, χαμηλή κύρωση. Όταν όμως ε, έχουμε ε, πλήρη ακύρωση της δραστηριότητας, όπως ας πούμε αναφέρθηκε για την μπανάνα ή όταν κάποια μέτρα θα καταδικάσουν ολόκληρες περιφέρειες και ολόκληρες παραγωγές, τότε δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για αντισταθμιστικά μέτρα, γιατί τι είδους αντισταθμιστικά μέτρα θα είναι αυτά. Η Ευρώπη δεν θα έχει αρκετά χρήματα έτσι ώστε να προχωρήσει σε τέτοιες αντισταθμίσεις, ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές όπου καλύπτονται ε, μονάχα από μία παραγωγή. Ορισμένα πράγματα να πω λοιπόν. Πρώτον, το να αναλύσει κανείς ένα ε, προϊόν στην εισαγωγή του ε, στο ευρωπαϊκό ε, χώρο δεν είναι το ίδιο με τον έλεγχο όλης της αλυσίδας παραγωγής του και θα συμφωνήσω ε, με τα ευρωπαϊκά όργανα τα οποία ε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δηλαδή, ε, ένας δειγματοληπτικός έλεγχος στην εισαγωγή δεν ισοδυναμεί με έλεγχο της παραγωγής. Δεύτερον, πριν από μερικούς μήνες είχαμε θυελώδεις συζητήσεις για την προετοιμασία της Κοπενχάγης ασχοληθήκαμε με μεγάλη ανησυχία για το μέλλον του πλανήτη, για την αποψήλωση των δασών, την επερήμωση κλπ. Ε, όμως βλέπουμε ότι στην ουσία έκτοτε έγιναν ακόμα πιο εκτατικές οι καλλιέργειες και πιο εντατικές. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα τμήματα των δασών του Ισημερινού αποψηλώνονται, καταστρέφονται έτσι ώστε να δημιουργηθούν ε, καλλιεργήσιμες γέες. Άρα αντί να πηγαίνουμε καλύτερα πηγαίνουμε χειρότερα. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες παραγωγής ε, στις χώρες αυτές. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται στις χώρες αυτές και όταν οι ίδιες ε, οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών καταδικάζουν τους τρόπους παραγωγής ε, όταν ας πούμε στην Βραζιλία η, ε, η υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία της υγείας και τον έλεγχο υγιεινής ε, της γεωργικής παραγωγής καταγγέλει τρόπους παραγωγής τότε δεν είναι δυνατόν αυτού του είδους ε, ε, οι παραγωγές και τα προϊόντα να γίνονται δεκτά από την Ευρώπη. Και σύμφωνα με την έκθεση στην οποία αναφέρομαι, ούτε για την Κίνα δεν είναι καλά τα προϊόντα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Μισελ Χάρκιν και μετά η Ελιζαμπέτ Γκέγκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Παπαστάμκο, για τα σχόλια που μας έκανε και περιμένουμε την έκθεση και περιμένουμε και τη συνεργασία μαζί του. Ε, εν συντομία θα ήθελα να σχολιάσω για τη συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο για την ε, Μερκοσούρ και συμφωνώ με πολλούς προλαλήσαντες ότι έδειξε αλαζονή η Επιτροπή στον τρόπο με τον οποίο απάντησε στους ευρωβουλευτές ε, και λίγο αργότερα εγώ έκανα μια συνάντηση με τον Επίτροπο λίγο μετά το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων και μου είπε απευθείας ότι αν θέλουμε να έχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία θα πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις στη Γεωργία. Αυτό έγινε πριν αρχίσουν καν οι διαπραγματεύσει. Και το είπε ο Επίτροπο πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Και συμφωνώ με τον τελευταίο ομιλητή που είπε ότι μερικέ φορέ η γεωργία είναι το μόνο αντάλλαγμα το οποίο δίνουμε για παραχωρήσει. Και ε, δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσει και θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Και νομίζω ότι ε, ε, δυσκολεύει και το κλείσιμο του γύρου της Ντόχα, αυτή τη συζήτηση που κάναμε σε σχέση με τη Μερκοσούρ. Και μιας και μιλήσαμε για το γύρο της ε, Ντόχα, θα είπα ότι φαίνεται ότι αφήνουμε κάποια παραχώρηση στο Βόλιο Κρέας και πρέπει να ξαναδώσουμε κάποια παραχώρηση στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Και θα πρέπει να δούμε τι παραχωρήσεις τελικά και τι δεσμεύσεις έχουμε. Εμείς ε, ως Επιτροπή θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τον προϋπολογισμό που έχουμε για τη Γεωργία σύμφωνα με ε, τις προοπτικές μέχρι το 2013 και θα πρέπει να δούμε και σε σχέση με τις συμφωνίες, με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών να δούμε τι ανταλλάγματα μπορούν να δοθούν. Οι Γεωργοί δεν θέλουν αντιστάθμισμα, θέλουν να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν και θα πρέπει να διαχωρίσουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε να, να, να μην τα εξετάζουμε χωριστά, αλλά αντιθέτως να τα εξετάζουμε σαν δέσμη μέτρων. Και συμφωνώ και με τον κύριο Καπούλα ε, Σάντο ότι θα πρέπει ε, να κάνουμε μια σωστή συζήτηση, να υποστηρίξουμε το ελεύθερο εμπόριο, αλλά να μην το αφήνουμε στην αγορά, γιατί δεν θα υποστηρίξει η αγορά τη γεωργία. Θέματα προτύπων, θέματα ποιότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι κομμάτι του γεωργικού μοντέλου στην Ευρώπη. Και εμεί ω Επιτροπή Γεωργία πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αν δεν τα προστατεύσουμε εμεί, θα χαθούν. Μια τελευταία σκέψη τώρα. Θυμάμαι όταν έγινε η συζήτηση για το REACH, όταν ήταν πριν από δύο χρόνια επίκαιρη συζήτηση για το REACH, κάποιος συνάδελφος, που, η κυρία Εκ, που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό, και εγώ είχα επιστολέ από μικρέ επιχειρήσει από κάποιου που πίστευαν ότι θα φυγούν από τη Ρίτς και το συζητούσα με την κυρία Εκ και μου είπε η κυρία Εκ ότι κάποια στιγμή όλα τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ενταχθούν σε αυτέ τι διατάξει για τη Ρίτς. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το, την ίδια οπτική γωνία. Δηλαδή όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν αντίστοιχα στάνταρτ σε σχέση με αυτά τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Χάρκιν, η κυρία Ελίζαβετ Γέγλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον συνάδελφο τον κύριο Παπαστάμκο και όλους τους συναδέλφους που υποστηρίζουν αυτά που μας είπε ο κύριος Παπαστάμκος. και οι πράσινοι και ο κ. Χόσλινγκ είχαν διαφορετική άποψη για τη δική μου ε, έκθεση, αλλά χαίρομαι που υποστηρίζουν τον κύριο Παπαστάμκο σε αυτό. Ήμουν, είχα πάει στον Καναδά με την αντιπροσωπεία και είχα τη δυνατότητα να πάω σε τρει επαρχίε και να μιλήσω με τρει ε, υπουργού γεωργία στι τρει περιφέρειε. Και οι τρει υπουργοί γεωργία ε, μου είπαν ότι έχουμε μια διμερή συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε με τον Καναδά αυτή τη στιγμή. Μου είπαν και οι τρει αρμόδιοι υπουργοί ε, ότι και βέβαια θέλουμε την εσωτερική αγορά της Ευρώπης για τα προϊόντα μας. Αλλά για ορισμένα προϊόντα όπως το γάλα, παραδείγματος χάρη, η δική μας αγορά παραμένει κλειστή. Ε, ε, ε παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά πιο δύσκολη. Και εγώ τους είπα πώς είναι δυνατόν ε, να γίνεται αυτό, γιατί οι Καναδοί καταναλωτές επωφελούνται από αυτά τα προϊόντα. Και με αντίστοιχε συμφωνίε θα μπορούν να υποφεληθούν και άλλε χώρε ολόκληρο τον κόσμο και θα ήταν ενδιαφέρουσα κανονικά και η ευρωπαϊκή αγορά. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε εμείς ε, πράγματα τα οποία ε, δεν επιτρέπουν άλλοι στις αγορές τους. Και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι ε, να ε, ενώσουμε τη φωνή μας για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το οποίο είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Συμφωνώ με όλους ότι δεν θέλουμε προστατευτισμό για το μέλλον. Ούτε το θέλουμε, ούτε το χρειαζόμαστε. Αλλά η οδηγία ρίξη ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα δεν μπορούμε να δεχτούμε το να μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει ολόκληρος ο κόσμος να δεχθεί τη δική μας νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Μπορεί να ισχύσει για μας, αλλά να μην προσπαθούμε να γενικεύσουμε τα πάντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση και θα πρέπει ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να δουν ότι εμείς είμαστε μια Επιτροπή Γεωργίας που δεν προσπαθεί να προστατεύσει τους γεωργούς της Ευρώπης, αλλά προσπαθούμε ε, να προστατεύσουμε το βιωτικό μας επίπεδο στην Ευρώπη. Έχουμε κάποια πρότυπα τα οποία είναι τα πρότυπα των δικών μας των καταναλωτών. Και να μην αφήσουμε μόνο την καναδική κυβέρνηση να υπερασπίζει τα συμφέροντα των δικών της καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ελίζαμπετ. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Κύριο Γιάκ, ε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία ε, είπαν και προηγούμενοι ομιλητέ. Τα είπε και η κυρία Μαγκίνε αυτά που ήθελα να πω. Και όλοι συμφωνούμε όσον αφορά τα προβλήματα της γεωργίας. Συζητήσαμε στην Ολομέλεια τα θέματα της Μερκοσούρ και είδαμε ότι υπάρχουν ανεπαρκείς διατάξεις και δεν μπορούν να συνεχίσουν τέτοιες διατάξεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαστάμκο για την έκθεση που μας ε, παρουσίασε. Θα πρέπει να βρούμε ε, ε, τα στοιχεία τα οποία ε, από κοινού με άλλες αρμόδιες επιτροπές θα προωθήσουμε. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτά τα θέματα, θα συνεργαστούμε με άλλες επιτροπές. Όταν μιλάμε για εισαγωγέ αυτοκινήτων, δεν θα αφήναμε να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκίνητα με προβλήματα στο σύστημα πέδησης, παραδείγματο χάρη. Αντίστοιχα, θα πρέπει να έχουμε κάποια πρότυπα και για τον τομέα της γεωργία και για τα γεωργικά προϊόντα και νομίζω ότι θα πρέπει και το Κοινοβούλιο αλλά και η Επιτροπή να συμφωνήσουν από αυτού. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όταν θα συνεδριάσουν οι συντονιστές για αυτά τα θέματα να δουν και το τι θα κάνουμε με τη Μερκοσούρ και τι θα κάνουμε και με τις ερωτήσεις της ε, κυρίας Μαγκίνες, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να δούμε τι δεν μπορεί να συνεχιστεί και τι πρέπει να αλλάξουμε στο μέλλον. Βεβαίως και είμαστε υπέρ του ελεύθερου και δικαίου εμπορίου, αλλά θα πρέπει σαφώς ε, να παρέχουμε τις διασφαλίσεις για όλους τους κλάδους, όχι μόνο για τη βιομηχανία, για όλους τους κλάδους και θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τους αντίστοιχους ε, συναδέλφους σε άλλες επιτροπές. Εύχομαι καλή, τύχη στον, καλή επιτυχία στον κύριο Παπαστάμκο για την έκθεση αυτή και όλοι θα περιμένουμε ε, τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης. Ευχαριστούμε. η Επιτροπή Εμπορίου συνδέεται με την ε, δική μας και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία με τον κύριο Παπαστάμκο, τον εισηγητή μας, θα είναι εξαιρετική. Ο κύριος Μποβέ έχει το λόγο. Καλημέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη άφηξή μου, αλλά ε, υπήρξαν προβλήματα με τα δρομολόγια των τρένων και των αεροπλάνων και δυστυχώς δεν μπόρεσα να φτάσω έγκαιρα. Πολύ σύντομα δύο-τρία πράγματα ε, και ελπίζω δεν θα, δεν θα ε, πω τα ίδια πράγματα, δεν θα επαναλάβω πράγματα που έχετε πει ήδη. Όταν μιλάμε για διεθνές ε, εμπόριο, να θυμόμαστε όλα αυτά που έχουμε πει στην Επιτροπή Γεωργίας, ε, δηλαδή ε, η, ε, η δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τις κερδοσκοπικές αγορές. Δεν πρόκειται να υπάρξει σωστή γεωργική πολιτική αν δεν καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία των γεωργικών αγορών. Νομίζω ότι η διασύνδεση είναι σαφής. Για να έχουμε μία σωστή αγορά θα πρέπει να βγάλουμε την κερδοσκοπία απ' έξω. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να με ένα ερώτημα. Σήμερα ε, ξέρουμε τη δομή των διεθνών αγορών ε, και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, ε ορισμένες επιχειρήσεις συγκεκριμένες οι οποίες ελέγχουν η Cargill, η Louis Dreyfus, η EDM, τέσσερις στην ουσία που ελέγχουν τους σπόρους και μάλιστα με διαδικασίες απολύτως αδιαφανείς όσον αφορά τη λειτουργία των εταιριών, όσον αφορά ε, τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν στις εμπορικές τους πρακτικές. Η καργίλα, ας πούμε, ε, δεν ξέρουμε καν από πού προέρχονται οι σπόροι της, ούτε καν τι είδους οργάνωση έχει ε, στην επιχείρησή της. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει πολύ σωστή δουλειά με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να να ε, μιλήσουμε, να αντιμετωπίσουμε μάλλον το πρόβλημα αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων. Όχι δηλαδή το πρόβλημα αναχώρα, αλλά αυτό το, το, το μεγάλο πρόβλημα των επιχειρήσεων. Τρίτον, επανήλθαμε ε, στη Συμφωνία Ευρώπη-Μερκοσούρ και ε, στη διάρκεια της ε, συζήτησης αναφέρθηκα σε ένα κατά την άποψή μου πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όπως είπε και ο Μισελ Νταντέν προηγουμένως όσον αφορά αυτήν την υπηρεσία υγεία. το θέμα της εταιρεία Tyson που είναι το νούμερο ένα των πουλερικών στον κόσμο. Στην τελευταία λοιπόν έκθεση αναφέρεται σαφώς ότι θα θα δημιουργήσουμε τρεις ε, ε, μονάδες στη Βραζιλία έτσι ώστε να δημιουργήσουμε γέφυρα εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν τους ενδιαφέρει να εγκατασταθούν στη Βραζιλία γιατί τους ενδιαφέρει η βραζιλιάνικη αγορά αλλά γιατί τους ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή αγορά. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Ε, είναι ανόητοι αν νομίζουν ότι θα είμαστε διαρκώς αφελείς. Και ε, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τις χώρες Μερκοσούρ σαν εφαλτήριο για να φτάσουν στην Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να ξαναδούμε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις εξαγωγών και νομίζω ότι αυτό θα σχετιστεί και με την γενικότερη συζήτηση για την ΚΑΠ. Επίσης, και εδώ ξανααναφέρομαι στην κερδοσκοπία, ε, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι έχει κάνει η Ευρώπη ε, όσον αφορά την ε, πολιτική βοήθεια προς τις λιγότερο ευνοημένες χώρες, τα πάντα εκτός από όπλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες ε, οι οποίες ακόμα και αν αναπτύξουν την αγορά τους θα κατακρινιστούν οι τιμές και επομένως ε, η κατάσταση θα είναι εξίσου τραγική. Θα πρέπει να έχουμε συνεργασία με χώρες, μια λογική συνεργασία και όχι μια λογική σαν αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Θα δώσουμε τώρα τον ε, λόγο στους εκπροσώπους, μάλλον στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί βλέπω ότι δεν ε, υπάρχει κάποιος άλλος από την Επιτροπή μας. Θα ήθελα καταρχήν να υπογραμμίσω τη συμφωνία αυτής τη έκθεση. Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί το εμπόριο είναι ένα δυναμικό στοιχείο για την αύξηση του, της ε, ανάπτυξης, παγκόσμιας ανάπτυξης εδώ και πολλές δεκαετίες. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια σημαντική μείωση του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου. Όπως το είπε και ο κ. Παπαστάμικος, συνολικά συρρυκνώθηκε κατά 12% το παγκόσμιο εμπόριο. Το 3% όμως, ε, στο 3% όμως ήταν η μείωση ε, του γεωρικού εμπορίου. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι σε ό,τι φορά τις εξαγωγές μας, όπως είπε ο κ. Παπαστάμικος, Μαζί με τις ΗΠΑ είμαστε η βασική εξαγωγή του κόσμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός παίκτη στο γεωρικό εμπόριο στον κόσμο. Κατά μέσο όρο, 2007-2009 οι εξαγωγές μας σε δολάρια ήταν 108 δισεκατομμύρια δολάρια. 107 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν εξαγωγή των ΗΠΑ κατά μέσο όρο. Το 2009 104 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν οι δικέ μα εξαγωγέ και το ίδιο ακριβώ ποσό είχαν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν και οι, δύο σχηματισμοί, α πούμε, να το πω έτσι, ε, αντιπροσωπεύουμε κάτι λιγότερο από το, 18, από το 80% των εξαγών των ε, προϊόντων στον κόσμο. Ε, η Βραζιλία έχει αυξήσει πολύ τι εξαγωγέ τη έχει πολλαπλασιάσει επί 4 από το 1999-2001, από 14 δισεκατομμύρια, έχει φτάσει στα 55 δισεκατομμύρια. Είναι ο άλλος βασικός παίκτη στο παγκόσμιο εμπόριο γεωρικών προϊόντων. Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τι εισαγωγέ, είμαστε βέβαια ο μεγαλύτερο εισαγωγέας στον κόσμο. Αντιπροσωπεύουμε το 19 περίπου των παγκόσμιων εισαγωγών, τουλάχιστον το 2009, κατόπιν με 14% είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά η Κίνα για πρώτη φορά το 2009 τρίτος εισαγωγιάς στον κόσμο. Αν δούμε την ακροπρόθεσμη εικόνα του παγκόσμιου εμπορίου και, του, της, και ε, ε, της, ε, το πώς εξελίσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι για πολλά χρόνια είχαμε ένα μικρό έλλειμμα. Ένα έλλειμμα το οποίο όμως μειώνεται Το 2006 μάλιστα είχαμε και πλεόνασμα, σχεδόν και το 2007. όλα αυτά βέβαια άλλαξαν με την οικονομική κρίση. Το 2008-2009 δεν είναι χαρακτηριστικές χρονιές. Εξαιτίας ακριβώς της ε, σημαντικής αύξησης των τιμών το 2008 και τη σημαντικής μείωση το 2009. Όμω όπω είπε και ο κύριος Παπαστάμκο, το σημαντικό είναι ότι εξάγουμε τελειοποιημένα προϊόντα, τελικά προϊόντα υψηλή ε, αξία, ε, κρασία αλκοολούχα προϊόντα, ε, μεταποιημένα προϊόντα, τρόφιμα. 12 από τα, πιο, τα 15 προϊόντα πιο πολύ εξάγουμε είναι τελικά προϊόντα. Και γι' αυτό το λόγο και οι βασικοί μας πελάτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, που έχει φτάσει στη δεύτερη θέση των πελατών μας τελευταία χρόνια, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Νορβηγία και τελευταία η Κίνα. Με την αύξηση των καταναλωτών που μπορούν να αγοράζουν τέτοιου είδους προϊόντα υψηλή αξίας Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές εισάγουμε κυρίως πρώτε ύλε, ε, τροφές ε, και κοσμένα τροπικά προϊόντα, κακάο, καφέ, μπανάνε, που τις Περισσότερε φορέ χρησιμοποιούμε σε προϊόντα τα οποία αργότερα θα εξάγουμε. Ή, εν πάση περιπτώσει, σε προϊόντα υψηλή αξίας. Μόνο έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε τις εξαγωγές μας και να μειώσουμε το έλλειμμά μα να το κάνουμε πλεόνασμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Λοιπόν, το βασικό χαρακτηριστικό του, της εμπορικής μας ε, κατάστασης στον κόσμο είναι ότι οι εισαγωγές μας είναι πρώτες ή τελικά τροπικά προϊόντα που έρχονται κατά 75% από τροπικές χώρες. Κατά 72% από τροπικές χώρες. Αυτές οι εισαγωγέ είναι απαραίτητες για να παρασκευάσουμε εμείς τελικά προϊόντα υψηλή αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαγωγέ μα είναι τέτοιου είδου προϊόντα ε, που εξάγονται σε σχετικά πλούσιους καταναλωτές. Οπότε η υψηλή ποιότητα χαρακτηρίζει την παραγωγή μας. Και αυτό το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Τα ευρωπαϊκά τυριά, το ευρωπαϊκό ζαμπόν, το ευρωπαϊκό κρασί ε, είναι τα καλύτερα και αυτά που πιο πολύ προτιμούν οι παγκόσμιοι καταναλωτές που αντέχουν να τα αγοράσουν. Συνεπώς, υψηλή ποιότητα, ε, έξυπνη λειτουργία της ε, αγοράς και ποιοτικές εταιρείε είναι τα βασικά μα χαρακτηριστικά για να προωθήσουμε τις εξαγωγές μας. Όμως, για να περάσω και ένα μήνυμα σε σχέση με τις πολυμερεί και τις διμερείς συμφωνίες που διεξάγονται, να πω το εξή. Τα, η ποιότητα των προϊόντων μας είναι στο κέντρο των ανησυχιών μας. Και γι' αυτό το λόγο πάντοτε τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνουμε τι γεωγραφικέ ενδείξει στα ε, προϊόντα για τα οποία διαπραγματευόμαστε. Και στις διμερείς και στις πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες διαπραγματευόμαστε. Θα ήθελα να σας πω ότι και εμείς ως Κομισιόν και ως Γενική Διεύθυνση ε, Γεωργίας ε, είμαστε πρόθυμοι να σας δώσουμε οποιασδήποτε πληροφορίε χρειάζεστε για να σας ε, βοηθήσουμε στην επεξεργασία αυτή τη έκθεση. Όχι όμω μόνο για αυτή την έκθεση. Οποτεδήποτε μας χρειάζεστε σε οποιαδήποτε συζήτηση θέλετε να διεξάγετε για θέματα διμερών ή πολυμερών ε, συμφων, εμπορικών συμφωνιών, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Molto bene. Ευχαριστούμε πολύ και τον Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως ε, Γεωργίας και θα δώσω τώρα βεβαίως το λόγο στον συνάδελφο κύριο Παπαστάμκο έτσι ώστε να εξάγει κάποια ε, συμπεράσματα και μετά να προχωρήσουμε με τη μέση διάταξή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Νικηφόρο Σιβένα να τον ευχαριστήσω για την ε, συνεισφορά του στη δική μας συζήτηση και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι θα συνεργαστούμε ε, γιατί ο κύριος Σιβένας εμφανίστηκε εδώ ε, πλήρως πεπισμένος για την ανάγκη ε, μιας, μάλλον ως φορέας μιας νέας διαθεσμικής κουλτούρας μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτή απορρέει και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και θέλω να πω επίσης ότι οι συνάδελφοι, αλλά και ο Μιλών, όσα είπαμε για την Επιτροπή, δεν αφορούν ε, την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, αλλά αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον κύριο Μποβέ και ιδιαίτερα συγκράτησα τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις κερδοσκοπικές αγορές αλλά και αυτό που είπε ότι οι χώρες Μερκοσούρ χρησιμοποιούνται ως εφαλτήριο για εξαγωγές ε, προς την Ευρώπη όπως επίσης για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας Everything But Arms ε, σε ό,τι αφορά τις αγωγές από ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ε, ε, ειδικά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Γιάρ ε, σε ό,τι αφορά τις αγωγές αυτοκινήτων, γιατί τα προβλήματα που μπορούν να εμφανίζουν αυτές τις αγωγές και την άμεση αντίδραση που έχουμε. Βεβαίως και τις αγωγές αυτοκινήτων και τα αυτοκίνητα και τα προβλήματά τους συνδέονται με την ασφάλεια των όλων ημών των οδηγών, αλλά και οι εισαγωγέ γεωργικών προϊόντων συνδέονται με την προστασία των καταναλωτών και με τη δημόσια υγεία. Συγκράτησα επίσης τις συνεισφορές της κυρίας Χάρκιν ε, και ιδιαίτερα ε, αυτό που είπε για το, για το σε ό,τι αφορά αν θα μπορούσαμε δεν δηλαδή να έχουμε ε, ένα ριτς για τις αγωγές γεωργικών προϊόντων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νταντέν, ο οποίο αναφέρει και στους τρόπους παραγωγής αλλά και στο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και ο οποίος ειλικρινά δούλεψε πάρα πολύ και αυτός μαζί στην προηγούμενη έκθεση την οποία κάναμε για την ε, ε, ΚΑΠ μετά το 2013, στον κύριο Μάτο, σε ό,τι αφορά το εύρος των διαπραγματεύσεων υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την κυρία Γκέγκλε και αυτή την εμπειρία που μας μετέφερε από το πώς λειτουργεί ε, και πώς αντιδρά ο Καναδάς σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ε, ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων τις δικές τους εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μεταφέρει και ως ατμόσφαιρα ε, αυτό το οποίο βίωσε η ίδια κατά τις επαφές με ε, Καναδούς αξιωματούχους την κυρία Χέραντς Γκαρσία και ιδιαίτερα ότι πράγματι οι αγρότες αγνοούν τις πιέσεις που που προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δεν είναι εξοικειωμένοι. Και οι, και οι οργανώσεις των αγροτών με αυτές τις επιπτώσεις και, και οι καταναλωτές, όχι μόνο η Ευρώπη, οι, Ευρώπη, οι αγρότες. Ε, με τον κύριο Νίκολσον ε, έχει αποχωρήσει, αλλά ε, τα είπαμε σε ό,τι αφορά τη στάση ε, του Επιτρόπου και ιδιαίτερα θέλω να συγκρατώ τις Παρατηρήσει του για τι ψηλέ προδιαγραφέ, την ισοδυναμία δηλαδή προδιαγραφών, τον κύριο Χόισλινγκ ε, με, σχετικά με τι διαπραγματεύσει, τα αποτελέσματα με τι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε που να έχουμε και να τονιστούν κατά τι διαπραγματεύσει με τρίτες χώρε τα προβλήματα των ε, Ευρωπαίων Γεωργών για τις διαπραγματεύσει συμφωνιών με τρίτε χώρε, και αυτό που το οποίο είπε ότι πρέπει να διασφαλίσει, το συνάδελφοι, το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και σε αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Λεφόρ, δηλαδή στην ασυμμετρία παραχωρήσεων μεταξύ γεωργικών προϊόντων και βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων πολυμερών ή διμερών με τρίτες χώρες ή ομάδων χωρών. Και ο κύριος Ντές αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό μοντέλο, που πρέπει να συνυπολογιστεί στις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες, όπως και ο κύριο Λαβία σε ανταγωνιστικότητα των δικών μας παραγωγών και πρέπει να σεβαστούμε τις πιέσεις που δέχονται οι δικοί μας παραγωγοί και ιδιαίτερα συγκράτησα και την παράμετρο του κοινωνικού ντάμπινγκ το οποίο έθεσε που μαζί βεβαίως με το οικολογικό ντάμπινγκ είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Και θα ήθελα να διαβιώσω τον κύριο Καπούλα Σάντος ότι ε, προσωπικά δεν είμαι υπέρ ε, μιας ε, βολονταριστικής προσέγγισης ή ενός ευχολογίου το οποίο θα πρέπει να απευθύνουμε στους Ευρωπαίους αγρότες υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης. Ε, έχω πλήρη συνείδηση και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έναντι τρίτων χωρών ε, και του ανοίγματο το οποίο έχει προβεί και βεβαίω είμαστε κατά του προστατευτισμού αλλά από την άλλη ότι θέλουμε ένα ελεύθερο πλην όμως δίκαιο ισορροπημένο εμπόριο αυτή είναι η πραγματικότητα και ε, προσβλέπω και στη στενή μας ε, συνεργασία. Και ευίωσα τα όσα είπε η κυρία Μαγκίνες ε, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εύλογη αντίδρασή της και θα ήθελα να πω ότι όταν συζητιέται ένα θέμα το οποίο άπτε των δικών μας αντικειμένων εδώ στην Ολομέλεια θα μπορούσαμε κύριε Πρόεδρε τουλάχιστον στη διαδικασία του Catch να δίνετε προτεραιότητα στους συναδέλφους που προέρχονται από την Επιτροπή Γεωργίας και όχι, και αυτό αφορά το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και όχι προς συναδέλφους ε, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με, το, με την Επιτροπή Γεωργίας, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Ωραία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους για την εξαιρετική ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχηθούμε βεβαίως καλό κουράγιο ε, στον εισηγητή κύριο Παπαστάμκο. Και φτάνουμε στο σημείο 6 τη ημερησία διατάξεω. Θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2011, έτσι όπω τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, το Συμβούλιο θα προτείνει σημαντική μείωση των γεωργικών γραμμών του προϋπολογισμού. Η πρόταση που ε, θα επιβεβαιωθεί ενδεχομένως στο Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου, αύριο δηλαδή, προβλέπει μείωση 811 821 εκατομμυρίων ε, και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Θα ήθελα να πω σχετικά με την έκθεση αυτή, να το πω σε όλους τους συναδέλφους, ότι ε, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών για την έκθεση αυτή, λέγω, είναι η 16 Ιουλίου, 12 το ε, μεσημέρι. Και θα δώσω αμέσως το λόγο, λοιπόν, στην συνάδελφο Μάιρετ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για να συνεχίσω από εκεί που μείναμε στο προηγούμενο θέμα, εάν θέλουμε ε, αντισταθμίσεις, να προβλέψουμε αντισταθμίσεις για όλα τα προβλήματα ε, των γραμμών του προϋπολογισμού, τότε σίγουρα δεν θα φτάσουν τα χρήματα. Διαδικαστικά τώρα, είπατε κύριε Πρόεδρε ότι αύριο θα έχουμε αποσαφηνήσει ε, όσον αφορά το, την, τις, προ, τις ε, στην προηγούμενη εβδομάδα όμως είχαμε μια συζήτηση ε, και με τον εισηγητή για τον ε, προϋπολογισμό και νομίζω ότι ακούσαμε πολλά πράγματα τούτη τη στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πολύ κοντά την διαδικασία και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δουλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια όσον αφορά τα αριθμητικά, τα αριθμητικά στοιχεία γιατί δεν είναι καθόλου ικανοποιητική η πρόσβαση που έχει το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του Κοινοβουλίου ε, στα αριθμητικά ε, στοιχεία. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αμεσότερα την πληροφόρηση από το Συμβούλιο και όχι να φτάνει μέσω των εκπροσώπων του τύπου η πληροφόρηση σε εμάς. Μέση λοιπόν πληροφόρηση από το Συμβούλιο. Και Ε, φαίνεται ε, σε αυτή την ε, περίπτωση ότι η θέση που παίρνει το Συμβούλιο είναι λίγο διαφορετική, δηλαδή στοχεύουν κάποιες, σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να μας πει δύο λόγια σχετικά με αυτόν τον ε, μηχανισμό to this, um, συμψηφισμού των ε, λογαριασμών. Ε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε από τον Γενικό Εισηγητή ότι γίνεται μια προσπάθεια να θεωρηθεί η γεωργία σαν ένα μεγάλο αποθεματικό από το οποίο μπορούν ε, να ε, ε, βγαίνουν διάφορα κονδύλια. Αυτά θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Επίσης, παρεμβάσεις ε, για πρώτες ύλε. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, μας απασχολεί ε, και επομένως θα πρέπει να συζητηθεί και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Επίσης, ε, μείωση προβλέπεται στην γραμμή του προϋπολογισμού που προβλέπει κονδύλια για τους παραγωγούς. Εμείς συζητήσαμε το θέμα αυτό και είπαμε ότι θέλουμε να ενδυναμωθούν ακόμα περισσότερο οι οργανώσεις των παραγωγών και όχι το αντίθετο, και επομένως αυτές οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο δεν μας βρίσκουν καθόλου σύμφωνε. Επίση, η μείωση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ε, υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση της κοινή γεωργικής πολιτικής από το ευρύ κοινό, ε, αυτές, αυτή η περικοπή των κονδυλίων πάλι δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δούμε ε, πώς θα έχουν ακριβώς τα πράγματα. Και επίσης ε, μιλάμε εδώ για ένα περιθώριο το οποίο αρχικά θα έπρεπε να είναι 1,3 δις και τελικά έφτασε να είναι μόνο 852 εκατομμύρια. Για τον προϋπολογισμό του 2011 είχε γίνει πολλή συζήτηση όσον αφορά τα θέματα αυτά και η εξέλιξη των γεωργικών αγορών είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ε, και εάν έχει στη, στη διάθεσή της η Επιτροπή κάποιες ε, προβλέψεις ε, θα θέλαμε να τις έχουμε κι εμείς και επίσης εάν είναι δυνατόν να ενσωματωθεί κάποιο αποθεματικό στο, στις γραμμές αυτές έτσι ώστε η μεγάλη δυτικότητα που παρουσιάζουν και η μεγάλη εναλλαγή που παρουσιάζουν οι αγορές να μπορέσει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Η διακύμανση των τιμών είναι είναι πάρα πολύ μεγάλη τον τελευταίο καιρό και επομένως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντισταθμιστεί. Ε, όσον αφορά τώρα το θέμα της ε, υγείας ε, και όσον αφορά την προώθηση προγραμμάτων σχετικά με την καλύτερη υγιεινή της διατροφικής αλυσίδας, προβλέπονται κάποια προγράμματα τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν οπωσδήποτε. Εγώ θα προτείνω κάποιες τροπολογίες, προτείνω ας πούμε τη δημιουργία ειδική γραμμή του προπολογισμού για το γάλα, και άλλωστε και η συνάδελφος Γέγλε ε, πολύ έχει δραστηριοποιηθεί για το θέμα αυτό στο παρελθόν. Επίσης, ε, αναδιοργάνωση της βιομηχανίας και της παραγωγής κυρίως σε λιγότερο ευνοημένες ε, περιοχές, ενίσχυση των παραγωγών και των συνεταιρισμών. Αυτές, αυτά τα στοιχεία θα αναφερθούν στις τροπολογίες μου, θα αντιμετωπιστούν μάλλον ε, επίσης, όσον αφορά τη διακύμανση των τιμών, προτείνω να πάρουμε ε, χρήματα από, το, από τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν και να μπουν σε ένα αποθεματικό ε, και επίσης να υπάρξει δυνατότητα παρέμβαση όσον αφορά την, το γάλα και όσον αφορά και το βούτυρο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς κινείται η αγορά σε συγκεκριμένα προϊόντα. Ε, ειδικά σε αυτά τα προϊόντα μπορεί να κινηθεί πολύ άσχημα η αγορά και θα πρέπει να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, ε, ε, όλα αυτά τα μέτρα κτηνοτροφικά και και προστασίας ε, και εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική γραμμή 20 ε, εκατομμύρια ευρώ γιατί έχουμε προβλήματα ε, ασθενειών. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα αποθεματικό για να είμαστε πιο σίγουροι. 10 εκατομμύρια ευρώ τώρα προτείνουμε εμείς για τα δύο προγράμματα θέματα ε, ε, ε, προώθησης καλύτερων, ποιοτικότερων πρώτων υλών και ποιοτικότερης και πιο υγιεινής διατροφής. Επίσης, όσον αφορά αυτό το θέμα του, της των ε, λογαριασμών, ε, νομίζω ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά παρόλα αυτά εμείς ε, σαν, σαν Επιτροπή θα πρέπει να δούμε λίγο πόσα ακριβώς έχει ο προϋπολογισμός. Είναι πολύ θα πρέπει να δούμε, δηλαδή, ε, αν μπορούμε να δεχτούμε ένα τέτοιο υπολογισμό, γιατί οι κινήσεις που προτείνονται είναι οριακά απαράδεκτες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μεγκίνες. Ε, με μεγάλη προσοχή ακούσαμε την έκθεσή σας και καταλάβαμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να επιτύχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Έχω ένα σχόλιο, δεν ξέρω πώς άλλοι συνάδελφοι ήθελαν να μιλήσουν και να το θέσω εγώ αργότερα. Grazie onorevole adesso apriamo il dibattito, se qualcuno vuole... Ε, ωραία, να ξεκινήσει η συζήτηση. Αν δεν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, θα δώσω αμέσως το λόγο στην Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Γενικό Διευθυντή Μπότσμαν. Ο Τζοβάνι, ναι, Τζοβάνι, Τζοβάνι Λαβία. Διαφώτισέ μας, Τζοβάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πρέπει να πω ότι οι περικοπές των πληρωμών, έτσι όπως προτείνονται από το Συμβούλιο, οπωσδήποτε μας απασχολεί. Είναι ενσυχητική η περικοπή αυτή. Αλλά από αυτά που είπε η Μάιρεντ, σίγουρα πιο σύμφωνο με βρίσκει το θέμα της δημιουργίας αποθεματικού εν ώψη αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων της αγοράς. Επ' αυτού του θέματος πρέπει να συζητήσουμε οπωσδήποτε, αλλά μία δυνατή πρόταση πρέπει να την κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ακάλυπτους τους γεωργούς μας και να μην τους δώσουμε μία απαραίτητη στήριξη σε περίπτωση κρίσης. Επίσης θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το Συμβούλιο, ε, έκαναν ένα πρώτο, μια πρώτη επιλογή των ε, προγραμμάτων αυτών και έχουμε 21 προγράμματα που χαρακτηρίζονται ε, από το γράμμα α, δηλαδή προγράμματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και που μπορούν να προχωρήσουν με τη βοήθεια της Επιτροπής. Μεταξύ αυτών υπάρχουν ε, κάποια προγράμματα τα οποία αφορούν την Επιτροπή μας και επ' αυτών θα πρέπει να επιμείνουμε ειλικρινά για τα πιλωτικά αυτά προγράμματα, τουλάχιστον σε μία πρώτη φάση, θα έλεγα ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη πρικοδότηση από αυτή που αναφέρεται στο έγγραφο και μετά θα δούμε βεβαίως πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό ε, το αίτημά μας να αφορά αύξηση της χρηματοδότησης. Ε, κάτι διαφορετικό ε, είναι το Ταμείο του γάλακτος. Θα θυμάστε ότι εμείς είχαμε πάγιο αίτημα να γίνει το Ταμείο αυτό σταθερό. Όμως το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησαν το εργαλείο αυτό μεταβατικό και σχετικό με το προϋπολογισμό του 2010. Βεβαίως δεν λύσαμε το πρόβλημα του γάλακτος με τα 300 εκατομμύρια που δώσαμε ε, πέρσι και που δεν είμαστε καν σίγουροι ότι χρησιμοποιήθηκαν ε, κανονικά. Θα πρέπει όμως να στραφούμε προς το μέλλον, να δούμε το μέλλον και να δούμε κατά πόσον μπορούν να βρεθούν κάποια νέα εργαλεία για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του συγκεκριμένου τομέα, έτσι ώστε ο παραγωγικός κόσμος με μεγαλύτερη ηρεμία να ατενίζει το μέλλον. συμφωνώ με, την, ε, με το περιεχόμενο των προτινόμενων τροπολογιών σχετικά με την αύξηση των πιστώσεων. Ε, ενδεχομένως θα υποβάλω και εγώ κάποιες άλλες ε, τροπολογίες. Έχουμε όμως... Ε, έχουμε όμως ακόμα μέχρι τις 20 του μηνός περιθώριο και θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο Μεγκίνες. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Σμιτ. Uh, συγχαίρω την εισηγητρία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα και εγώ θα ήθελα να ζητήσω περισσότερες πληροφορίες. Ασφαλώς δεν είμαστε ε, η Επιτροπή των Προπολογισμών, αλλά έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαδικασία. Ιδιαίτερα, ε, δεδομένου ότι επέρχεται και το καινούριο καθεστώς της εποχής μετά το 2013. Πολλά θα αλλάξουν. Συνεπώς ε, και εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση για καλύτερη πληροφόρηση, περισσότερε πληροφορίε, Προτιμώ να μην διαβάζω τα πράγματα στις εφημερίδες ε, και ε, να τα ξέρουμε πριν μα τα θέσουν υπόψη μα οι ενώσει των παραγωγών ή τα συνδικαλιστικά του σε σωματεία. Οι περικοπές μας ανησυχούν. Θα υποβάλουμε και εμείς τροπολογίες ε, θέλω να πευθώ ε, το, στην Κομισιόν για το, για το παρατηρητήριο το οποίο πρότεινε η ομάδα των φιλελεύθερων. Πράγματι ε, είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά λειτουργεί σωστά. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε αντικειμενικά στοιχεία, με στοιχεία το πιλωτικό πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και κάποιο καιρό, αλλά δεν έχουμε δει αποτελέσματα. Συνεπώ, η Κομισιόν θα μπορούσε να μα ενημερώσει που βρίσκεται αυτό το στοιχείο, ε, αυτό το, αυτή η δραστηριότητα, αυτό το project. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη επίση για να διαθέτουμε πραγματικά αντικειμενικά στοιχεία για το κατά πόσο λειτουργεί η αγορά. Γιατί ενδεχομένω το project αυτό δεν κάνει αυτό το, για το οποίο προορίζεται. Ευχαριστώ. Grazie Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γέγκλε. Από την εμπειρία μου ω εισηγήτρια για τον προπολογισμό από πέρυσι, ξέρω πολύ καλά τι αντιμετωπίζει η Μέριν Μακίνες και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο. Και μου κάνει άλλη μια φορά εντύπωση η χαλαρότητα της Επιτροπής όταν λέει ότι με την απελευθέρωση υποφελείται η παγκόσμια αγορά και δεν θα χρειαζόμαστε τόσο πολλά χρήματα για την γεωργία. Δεν ισχύει και δεν θα ισχύσει ποτέ. Είναι υπεραπλούστευση κάτι τέτοιο. Πέρυσι είχαμε περισσότερα μέσα για τον, περισσότερους πόρους για τον προϋπολογισμό και πρέπει να το παλέψουμε και φέτος. Αλλά αυτό που χάνουμε είναι κάτι που έχει σχέση με την προοπτική του 2013. Γιατί ε, αν δεν μας δοθούν οι κατάλληλοι πόροι, θα επιδεινωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Και ευχαριστώ και τον Τζοβάνι για αυτά που είπε. και ευχαριστούμε για τις προσπάθειες, γιατί και εσύ και η Μακίνες ε, θα το παλεύσετε πολύ για να καταφέρουμε ε, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ και για όλα αυτά που είπαν άλλοι οι ομιλητές, αλλά πιστεύω ότι η απελευθέρωση δεν ταυτίζεται με καλύτερες ε, συνθήκες και προοπτικές για τους γεωργούς και είναι κάτι που το ακούσαμε και από την προηγούμενη έκθεση του κ. Παπαστάμκου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους εξίσωση. Θα πρέπει να δούμε ε, τα πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται και πώς αυτά έχουν επιπτώσει στον προϋπολογισμό. Σου εύχομαι πραγματικά καλό κουράγιο, Μέιριτ. Και σε, σε ευχαριστώ, Τζοβάνι. Λουίς Καπούλα Σάντος. Ε, η Μάργαρη πήρε τα λόγια από το στόμα μου. Ε, είναι και δικές μας οι ανησυχίες της κυρίας Μαγκίνες. Αυτό που πιο πολύ μας ανησυχεί όμως είναι η μείωση του προπολογισμού ε, και μείωση του περιθωρίου. η Κομισιόν είπε, είχε πει, ότι θα λάβει υπόψη τις ανάγκες για ένα αποθεματικό ε, μέσω, μιας, ε, μέσω ενός διορθωτικού προπολογισμού. Θα, ήθελα σε αυτό το θέμα η Κομισιόν να γίνει πιο σαφής. Ευχαριστώ. Grazie Luis, George. George, παρακαλώ. Ευχαριστούμε την κυρία Είμαι καινούριο σε αυτή την επιτροπή. Παρόλο που είμαι μέλος του Κοινοβουλίου εδώ και καιρό. Ε, εγώ σχολιάζομαι με τα οικονομικά του Σκοτσέζου Κοινοβουλίου παλιότερα. Θα ήθελα η λοιπόν να μου με ενημερώσει για το εξή. Μιλάμε για το προσχέδιο προπολογισμού του 2011. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως τα στοιχεία του φθινοπόρου, ε, διότι χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε προβλήσουμε το 2011. Αυτή τη ε, στιγμή η Κομισιόν προτείνει περικοπές με βάση ε, υποθέσεις που ενδεχομένως έχουν σχέση με την κρίση κλπ. Αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί η Κομισιόν και να περιμένουμε και το φθινόπωρο για να είμαστε σίγουροι. Επίσης θα πρέπει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι αν μειωθούν, να μειωθεί αυτό το προπολογισμό κατά αυτό το ποσό, τα χρήματα θα επιστραφούν στα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να εξοικονομηθούν από εδώ και να διατεθούν κάπου αλλού. 310 εκατομμύρια ευρώ είχαν κρατηθεί για την κρίση του γάλατος. Τώρα, αυτά τα χρήματα τελικά δεν δαπανήθηκαν. Ε, ποιο ήταν το πρόβλημα γι' αυτό ή δεν έχω καλή ενημέρωση, τι από τα δύο ισχύει. Το σε ό,τι αφορά τη συγκυρία. Σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών, όπως γνωρίζετε, γίνονται σημαντικές περικοπές δημόσιες δαπάνες. Και στη δική μου χώρα το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα κονδύλια που τα πανούμε και οποιαδήποτε, ε, οποιοδήποτε έτοιμά μας θα πρέπει να δικαιολογείται δεδομένης της οικονομικής συγκύρισης και των περικοπών σε εθνικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε και τον πραγματικό κόσμο στον οποίο ζούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, George. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τον ε, λόγο στην Κριστίνα Μπότσμαν ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ξέρω ότι βλέποντα τον προπολογισμό και αν δείτε την πρόταση της Επιτροπής και την πρόταση του Συμβουλίου για τις περικοπές, είναι πολύ τεχνικά όλα αυτά τα θέματα. Πριν απαντήσω λοιπόν σε κάποιες από τις ερωτήσεις και σχόλια, επιτρέψτε μου να εξηγήσω αυτή την καθάριση λογαριασμών ε, και όσον αφορά τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο. Δεν θα μιλήσω εγώ για την αιτιολόγηση των περικοπών, αλλά θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Έχουμε δύο διαφορετικά είδη καθάριση λογαριασμών. Έχουμε αυτά τα οποία γίνονται για λόγου συμβατότητα και αυτό είναι ω παράπλευρο έσοδο. Προτείνω αυτό να το αφήσουμε κατά μέρο, διότι δεν φαίνεται στον προπολογισμό. Αυτό το οποίο κάνει η Επιτροπή είναι ότι ε, υπολογίζει πώς είναι αυτά τα παράπλευρα έσοδα και τα μειώνει από τα αιτήματα πληρωμών. Επομένως, το καθαρό αίτημα στον προϋπολογισμό φαίνεται διαφορετικό. Παράλληλα, όμως, υπάρχει και η εκαθάριση λογαριασμών που είναι στο κεφάλαιο 0507, που είναι αυτό το οποίο λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη όταν κάνουν την ετήσια εκαθάριση λογαριασμών, αν ανεβρεθούν σφάλματα στους λογαριασμούς. Δεν μιλάμε για διόρθωση, μιλάμε για σφάλματα ή όταν τα κράτη-μέλη καθυστερούν πληρωμές. Οπότε και αυτό γίνεται έσοδο. Δεν είναι όμως παράπλευρο έσοδο, είναι έσοδο του προϋπολογισμού και αυτό ονομάζεται αρνητική δαπάνη. Το μέσο έσοδο σε αυτό το κεφάλαιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν 72 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό προτείνει η Επιτροπή στην πρότασή της να έχουμε έσοδα 72 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη γραμμή. Όμως το Συμβούλιο τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον πρότεινε να αυξηθεί αυτή η αρνητική δαπάνη. Αυτό γίνεται όχι διότι πιστεύει κανείς ότι θα έχουμε αυτό το έσοδο, απλώς διότι η Επιτροπή θα ήθελε να έχει λιγότερες δαπάνες σε όλα τα άλλα κεφάλαια που αφορούν τις ε, γεωργικές δαπάνες και στο τέλος του έτους όλες αυτές οι μικρότερες δαπάνες, οι μικρότερες δαπάνες να πάνε σε αυτή τη γραμμή και να κλείσουν αυτή την τρύπα. Γιατί δημιουργείται μια τρύπα από το Συμβούλιο την οποία πρέπει να κλείσει η Επιτροπή. Δεν θα το ερμηνεύσω εγώ το γιατί το Συμβούλιο επιλέγει αυτήν την τακτική, αλλά αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν θα πει ότι πρέπει να κάνουμε περικοπή σε αυτή ή σε εκείνη τη γραμμή. Λέει απλώ πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα δαπανίσει κάπου όλου στον προπολογισμό 420 εκατομμύρια λιγότερα και έτσι στα τέλη του έτου θα κλείσει αυτή η επιτροπη θα δαπανισει καπου αλλου στον προπολογισμο 420 εκατομμυρια λιγοτερα και ετσι στα τελη του ετου θα κλεισει αυτη η τρυπα Επανέρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο λέτε για την Επιτροπή, ότι είναι πολύ αισιόδοξη στις εκτιμήσεις της για τις δαπάνες των αγορών. Το είπα και πέρυσι που έρθει και θα το ξαναπώ τώρα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού είναι ρεαλιστικό, ούτω ώστε να μην έχουμε ένα προπολογισμό που να λέμε ε, θα είναι 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανών το 2011, όπως περιμέναμε ότι θα έχουμε και το 2010, γιατί μπορεί να υπάρξει και κάποια κρίση. αλλά αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι προτείνουμε ένα προπολογισμό με βάση την κατάσταση της αγοράς τη στιγμή που συντάσσεται ο προπολογισμό. Όμως έχουμε και την επιστολή τροποποίησης και μετά την συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να υπάρξει ε, επιστολή τροποποίηση από την Επιτροπή και θα υπάρξει και φέτο επιστολή τροποποίηση. και αυτό το οποίο θα ε, κάνει η Επιτροπή είναι ότι πριν από τη συνδιαλλαγή θα υποβάλει αυτή την, την επιστολή τροποποίηση και θα εξετάσει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάσταση τη αγορά. Η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού βέβαια θα το εξετάσει επίσης και προτείνω να μην βάλουμε κάτι σε αποθεματικό. Αν πάμε στο Συμβούλιο ή έρθουμε σε εσά και πούμε προσθέσαμε κάτι εδώ γιατί φοβηθήκαμε ότι θα υπάρξει κρίση, αυτό δεν θα οδηγήσει σε σωστό προπολογισμό. Αυτό το οποίο κάνουμε κάθε χρόνο είναι ότι φροντίζουμε να υπάρχει ένα περιθώριο. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται να υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε σε εσά αν υπάρχει κρίση και να ζητήσουμε με ένα τροποποιητικό προπολογισμό αυτά τα οποία χρειάζεται. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να, να, να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή κρίση. Δεν ε, είναι ρεαλιστικός τρόπος ε, της του προϋπολογισμού το να έχουμε αποθεματικό για κάποια κρίση. Προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκτίμηση και σας έχουμε στείλει ένα λεπτομερές έγγραφο εργασίας για φέτος με όλες τις ποσότητες, με όλες τις κλίμακες και όλες τις εκτιμήσεις της αγοράς. με την ε, μεταρρύθμιση του 2003 και με το health check της αγοράς έχουμε όλο και λιγότερες δαπάνες και έχουμε τις άμεσες ε, ενισχύσεις ε, πλέον. Και θα δείτε ότι φτάνουν οι άμεσες ενισχύσεις σχεδόν στο ανώτατο όριο. Για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έχουμε φτάσει στο 99% και δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη ε, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα οποία δεν είχαν δαπανίσει μέχρι τώρα για τα, τους πόρους του άρθρου 68. Υπάρχουν χρήματα λοιπόν, μόνο που δεν έχουν μπει αυτά τα χρήματα στο κομμάτι που αφορά τις αγορές. Τώρα όσον αφορά το Ταμείο για το Γάλα και τη μελλοντική προοπτική. Για φέτος έχουμε τη γραμμή 99 για τα 400 εκατομμύρια όσον αφορά το Ταμείο για το Γάλα και έχει δίκιο, δίκιο ο κύριος ότι δεν είχαμε πολλέ δαπάνε τον Απρίλιο, όμως είχαν προβλέψει τα κράτη-μέλη ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα είχαν δαπανίσει 295 εκατομμύρια. 10 Ιουλίου είναι η ημερομηνία αποστολή των δηλώσεων των κρατών μελών. Σήμερα δηλαδή λαμβάνουμε, σήμερα Δευτέρα, 12 Ιουλίου, θα λάβουμε τα στοιχεία που έστειλαν τα κράτη-μέλη και στις 20 Ιουλίου θα έχετε τα λεπτομερή στοιχεία ε, ακριβώς για το τι δαπανήθηκε και φαίνεται ότι πήγαν πολύ καλά τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, δαπάνη αυτών των χρημάτων. Περιμένετε όμω και θα τα δείτε τα στοιχεία αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα μελλοντικά στοιχεία, η κυρία Μακίνε είπε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για τη διαφοροποίηση και την αναδιάρθρωση. Διαφοροποίηση και αναδιάρθρωση είναι δύο μέτρα εξαιρετικά, τα οποία θα τα βρείτε στην ανάπτυξη τη υπαίθρου, όχι όμω στο τμήμα που αφορά τι αγορέ. Και επίση, υπενθυμίζω ότι το περσινό πακέτο ανάκαμψη επέτρεψε να δαπανηθούν πολλά χρήματα για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα. Και μάλιστα ήταν περίπου 300 εκατομμύρια που είχαν δοθεί και για τα προγράμματα ανάπτυξης από τα πακέτα αναδιάρθρωσης. Όταν θέλουμε κάτι στον τομέα των αγορών, θα πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα της ομάδας υψηλού επίπεδου. Αύριο το πρωί νομίζω θα το συζητήσετε με τον Γενικό μας Διευθυντή το θέμα του γάλακτος και της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου. Ο κ. Καπλεσάντος ρώτησε τι θα κάνει η Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων. Βεβαίως αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που θα πρέπει να συζητηθεί μετά το 2013. Και σίγουρα θα το συζητήσουμε. Και την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια ε, μεγάλη διάσκεψη με τον Επίτροπο, τον κύριο Τσούλος. Για ε, ε, το τι απέγινε το 2009 θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε 110 λιγότερες δεσμεύσεις ε, μετά τον τροποποιητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής. Ο τελευταίος τροποποιητικός προϋπολογισμός της Επιτροπής έδωσε 135 εκατομμύρια από τα αγροτικά μέτρα στο πακέτο της, της ε, ανάκαμψης και αυτό το οποίο απέμεινε ως δεσμεύσεις δαπανήθηκε από την Επιτροπή. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, υπήρξαν ε, λιγότερες δαπάνες, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμών ε, ε, επιστρέψαν πέρυσι για την αγροτική ανάπτυξη, γιατί υπήρξε κάποια επιβράδυνση μη αναμενόμενη λόγω τη κρίση, λόγω του γεγονότο ότι αναπρογραμ... αναπρογραμμάτισαν τα κράτη-μέλη λόγω ε, του, του health check και επειδή κάποια κράτη-μέλη καθυστέρησαν με τα προγράμματά του, είχαμε αυτή την υστέρηση. Αλλά η εκτίμησή μα είναι ότι το 2011 θα έχουμε αύξηση των δαπανών και θα φτάσουμε στι ίδιε δαπάνε, όπω και στα προηγούμενα έτη και ε, ε, γι' αυτό έχουμε βάλει ε, το ποσό αυτό για δαπάνη του χρόνου και πιστεύουμε ότι αυτό ε, θα τηρηθεί. Αν δεν έχουν μπει στην, ε, σε πλήρη ανάπτυξη των προγραμμάτων τα κράτη-μέλη και δεν δαπανίσουν τα συνολικά ποσά, ίσως έχουμε κάτι λιγότερο. Αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό για το 2012 και το 2013 και δεν έχουμε rollover στον ε, προπολογισμό της Επιτροπής, έχουμε αιτήσιο προπολογισμό, δεν μεταφέρουμε στον επόμενο. Αυτά τα οποία δεν δαπανώνται μπορούμε να πούμε ότι τα ε, δίνουμε πίσω στα κράτη-μέλη, αλλά μπορεί να πει κανείς ότι ποτέ δεν τα πήραμε από τα κράτη-μέλη, διότι δεν τα τραβήξαμε. Τα τραβάμε σιγά-σιγά όσο προχωρά η εκτέλεση του προπολογισμού. Υπάρχει μια δυνατότητα μεταφοράς ε, των πιστώσεων πληρωμών που δεν χρησιμοποιήθηκαν Είχαμε 600 εκατομμύρια για το, για το 2009, τα οποία μέχρι το Μάρτιο όμως είχαν προβλεφθεί. Επίσης, ε, για τις ε, δεσμεύσεις πληρωμών μπορούμε να έχουμε κάποια ε, μεταφορά και αυτό το είχαμε κάνει το 2008 Τελικά όμως έφτασε η κρίση και δεν δαπανίσαμε αυτά τα οποία είχαμε προβλέψει ότι θα δαπανίσουμε. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες, αλλά όχι για το Ταμείο Εγγυήσεων, γιατί εδώ έχουμε μη διαφοροποιημένες δαπάνες. Υπάρχουν οι δεσμεύσει που δεν δαπανώνται μέσα στη χρονιά μπορούν να δαπανηθούν την επόμενη χρονιά. Πάντω πέρυσι τα δαπανίσαμε όλα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για τις επεξηγήσεις και τις λεπτομέρειες που μας δώσατε, κυρία Κριστίνα Μπόσμαν. Μάιρετ, ξανά το λόγο σε σένα για να ολοκληρώσει τη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο για τα πιλωτικά προγράμματα, πιλωτικά σχέδια και μετά θα σχολιάσω τα, τις παρατήσεις των αντιπροσωπιών. Εμείς υποβάλαμε ως Επιτροπή στις δύο Ιουνίου στο ψήφισμά μας 7 τέτοια πληρωτικά προγράμματα. Πήραμε απάντηση για δύο από αυτά από την Κομισιόν. Ένα, για να ξαναρχίσουμε το πρόγραμμα για τη ε, διατήρηση της γενετικής ποικιλία στην ιδιωτική παραγωγή, ε, σπόρους και ε, λοιπά. Ε, υπάρχουν 17 σχετικές ε, μελέτες όμως, οπότε η Κομισιόν προτείνει να περιμένουμε ε, τέλος του επόμενου χρόνου θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματά τους με συστάσεις το 2012. Οπότε η Κομισιόν ζητά αυτό το πιλωτικό σχέδιο ε, να, ε, έχει, να εφαρμοστεί έτσι κι αλλιώς εξαιτίας των μελετών. Δεύτερο πιλωτικό πρόγραμμα για το οποίο πήραμε απάντηση σχετικό με τη δημιουργία ενός δικτύου για την ευζοία των ζώων. Η Κομισιόν είναι θετική και ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Η Κομισιόν έχει κρατήσει 14 εκατομμύρια για όλα τα πιλωτικά προγράμματα, έχει δεσμεύσει 14 εκατομμύρια και εδώ ακούω τον κύριο Λαβίρ. Πρότασή μας ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ να αποδοθεί σε καθένα από τα 7 σχέδιά μας. Ε, ε, αυτά που είχαν προτείνει δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση για τα πιλωτικά σχέδια. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τη διευκρίνηση σε ό,τι αφορά το λογιστικό ζήτημα. Όμως από ό,τι φαίνεται η ο, αυτό που κάνει το Συμβούλιο είναι φτιάχνει μια τρύπα και μετά ζητάει από τους άλλους να τη γεμίσουν. Η Κομισιόν θα αποφασίσει πώς θα τη γεμίσει, από πού θα κόψει δηλαδή να γεμίσει αυτή την τρύπα. Αυτό εμείς, που κάνουμε όμως εμείς ως Επιτροπή και μέσω των τροπολογιών και των προτάσεών μα είναι να προστατεύσουμε το γεωργικό τομέα και τον δικό του προπολογισμό. Οπότε, ε, ε, συμφωνώ με την κυρία Γέγκλα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος για τον γεωργικό προπολογισμό. Ο τομέας ήδη απειλείται και θα πρέπει να δούμε τι ψηφίσαμε στην ε, έκθεση Lion την περασμένη χρονιά για τον προπολογισμό, το γεωργικό προπολογισμό μετά το 2013. Αν επιτρέψουμε τώρα περικοπές, θα στείλουμε ένα πολύ αδύναμο μήνυμα. Ε, θα πρέπει να, είμαστε, να στείλουμε ένα πιο ισχυρό μήνυμα. Σε ό,τι αφορά τον Άλλα Σμιθ, Περιμένουμε τις τροπολογίες σας και τις προτάσεις σας. Συμφωνώ με το σχολείο σας. Δεν είναι χρήσιμο να παίρνουμε πληροφορίες από ομάδες πίεσης, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές. Θα πρέπει τις πληροφορίες να τις παίρνουμε κατευθείαν εμείς. Θα μπορούσαμε ίσως να οργανώσουμε και μια συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αυτό. Ίσως η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Ε, κ ε, θα λάβουμε υπόψη την προτάση σας. Ε, ε, τα 300 εκατομμύρια για το, του Ταμείου Γάλακτος έχουν ε, δαπανηθεί μάθαμε από την Κομισιόν, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε πώς ε, έχουν δαπανηθεί κάποια άλλη στιγμή. Επίσης δόθηκαν διευκρινήσεις για, για το ζήτημα του κατά πόσον ε, τα ποσά που δεν δαπανώνται επιστρέφονται στα κράτη-μέλη κλπ γνωρίζουμε ότι ο γεωρικός προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια ε, ε, είναι ε, αυτός ο οποίος απειλείται πιο πολύ οπότε, και θα απειλείται πιο πολύ, οπότε υπάρχουν ανάγκες. Θα προσπαθήσουμε με τροπολογίες να εξασφαλίσουμε ότι οι προτεραιότητές μας θα ξανατοποθετηθούν στο κέντρο της συζήτησης του προπολογισμού. Τροπολογίες λοιπόν μέχρι τις 20 Ιουλίου, μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ. Ωραία λέει ο Πρόεδρος. Το μόνο που πρέπει να προσθέσω είναι ότι ε, η προθεσμία υποβολής δεν είναι 20 Ιουλίου πλέον, ε, κυρία Μακγκίνες, αλλά η 16 Ιουλίου. Ε, γιατί για τεχνικούς λόγους έπρεπε να ε, θέσουμε σαν ε, χρονικό όριο για 16 Ιουλίου. Ελπίζω αυτό να μην σας προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για τις 16 Ιουλίου. Εάν τα καταφέρουμε έχει καλώς, γιατί διαφορετικά θα δώσουμε καμιά δυο μέρες ε, προθεσμία. Ε, παρακαλώ πολύ να θεωρήσετε ότι η 16 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι, είναι η τελευταία προθεσμία. Εκπνέει τότε η προθεσμία. Μια ερώτηση έχω. Αν πρόκειται για τις 16, είναι σχεδόν αδύνατο. 20 θα μπορούσε Αλλά να, να, μην έχουμε τόσο σύντομα τις προθεσμίες. Να μην βάζουμε τις προθεσμίες τόσο κοντά. Δεν τα καταφέρνουμε. Μάιριντ, Μακίνες. Ας είμαστε λίγο λογικοί. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να υποβληθούν σήμερα ή αύριο. Αν όμω κάποιοι συνάδελφοι ε, χρειάζονται περισσότερο χρόνο, να τους δώσουμε Είμαστε πολύ κοντά στις διακοπές όμως. Οπότε υποστηρίζω την ιδέα να καθορίσουμε την 16η Ιουλίου ως ε, ημέρα, ε, τελική ημερομηνία, για να ε, κάνουμε πιο γρήγορα τις μεταφράσεις. Αν τα καταφέρουμε αυτήν την ημερομηνία χωρί προβλήματα, α το προσπαθήσουμε. Τώρα εντάξει, αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα, να του δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Εγώ θα προσπαθούσα να περιοριστούμε στι 16 αν γίνεται. Ο George Lyon ζήτησε το λόγο. Για να συμφωνήσουμε πριν τη 16η, ίσως η ισω η κομισιον θα μπορούσε να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε ω ένα ενημερωτικό σημείωμα, για παράδειγμα. Ε, τι, πώς ε, κατανέμεται τα ε, ποσά ενίσχυση των αγορών στον προπολογισμό κλπ. Δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Τι, ποια περιμένουν θα είναι τα έσοδα από την πώληση αποθεμάτων παρέμβασης, τυριού, βουτύρου κλπ. που δημιουργήθηκαν τη διάρκεια της κρίσης του γάλακτος. Η Κομισιόν προβλέπει καθαρό κέρδος θα μπορούσε να μας υποβάλει ένα ενημερωτικό σημείο για το πότε θα πουληθούν, πώς θα πουληθούν κλπ. Γιατί ε, αυτό θα επηρεάσει τις γραμμές ε, του προβλησμού για την παρέμβαση του χρόνου. Ο λόγος στην Κομισιόν. Υπάρχει ένα έγγραφο εργασία ε, το οποίο το έχουμε στείλει στον πρόεδρο της Επιτροπής και ε, εξηγούμε με λεπτομέρειες όλα τα κέρδη τα οποία πιστεύουμε θα προκύψουν από την πώληση των αποθεμάτων. Ε, το διανύμαμε και στην ε, Επιτροπή Προπολογισμού. Σίγουρα θα προκύψει καθαρό κέρδος. Αυτή τη στιγμή πουλάμε βούτυρο από την παρέμβαση και με κέρδος. Και ε, το περισσότερο, ε, μεγαλύτερο κομμάτι του κέρδους θα καταλογιστεί στο 2010. Στην ε, επεξεργασία του προϋπολογισμού 2011 βέβαια δεν ξέραμε πότε θα πουλήσουμε το αποκορυφωμένο γαλαζοσκόνη κλπ. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τον προϋπολογισμό και θα υποβάλουμε βέβαια και ένα επεξηγηματικό έγγραφο για αυτές τις αναθεωρήσεις. Διμερώς θα συζητήσουμε για το άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Ωραία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μα ε, ζητούν ε, να σεβαστούμε την αρχική ημερομηνία τη 20 η Ιουλίου, ε, γιατί από ό,τι φαίνεται προβληματίζονται ιδιαίτερα, τότε, αγαπητή κυρία Μαγκίνες, να πούμε ότι εκπνέει η προθεσμία υποβολής τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι στις 20 Ιουλίου. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο νωρί, δεν τα καταφέραμε, τι να κάνουμε. Εάν ε, δεν υπάρχουν άλλες ε, αιτήσει για ομιλία. Να φτάσουμε στο σημείο 7, ανταλλαγή απόψεων με θέμα την εφαρμογή κανονισμού ΕΚ 21 2004 σχετικά με την ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η ομάδα του ΕΛΚ, μας ζήτησε να βάλουμε το θέμα αυτό στη μέση διάταξη. Από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με πληροφορίες, το εμπόριο προβάτων ανάμεσα στην Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδική Δημοκρατία αντιμετώπισε προβλήματα μετά από την εφαρμογή χωρίς πρώτερη συμφωνία κανόνων συγκεκριμένων όσον αφορά την ηλεκτρονική σήμανση. Παρακαλώ πολύ, ποιο θέλει τον λόγο. μιλάμε για την ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων, θέμα που βάλαμε στη μέση διάταξη μετά από αίτημα της δικιάς πολιτικής ομάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το θέμα αυτό, ο συνάδελφος ε, Πέτρο νομίζω ότι θα το έχει χειριστεί καλύτερα και προτείνω να του δώσουμε το λόγο. Εγώ, Γιάρ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα αφορά την ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων ε, και όποιος ε, είναι περισσότερα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξέρει ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών που αφορά, αφορούν ακριβώς ε, αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής σήμανσης που επειδή είναι πολύ γραφειοκρατικό γίνεται σχεδόν μη υλοποιήσιμο και ανέφικτο. Μπορεί να κοστίζει για τα βοηθή 100 ευρώ αναζώ και ε, είναι πάρα πολύ ε, υψηλή η δαπάνη για τα εγωπρόβατα και είναι σχεδόν ανέφικτο το σύστημα. Πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ε, μεταφέρει σε εθνική νομοθεσία και δεν έχουν εφαρμόσει αυτή τη διάταξη και υπάρχει πρόβλημα στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εκτροφείς προβάτων ε, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα λένε ότι αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τις διατάξεις ε, δεν είναι εφικτό. Ε, και πραγματικά να θέλει κανείς να, να, εφαρμόσει τις διατάξεις δεν θα τα καταφέρει. Θα μπορούσαν ε, ε, να οδηγηθούν και στην ε, εγκατάλειψη της δραστηριότητας και οι λύσεις τις οποίες έχουν δεν είναι βιώσιμες. Εμείς θέλουμε να έχουμε περιφερειακή παραγωγή και δεν θέλουμε να χάσουμε παραγωγούς προβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και με αυτό το σύστημα της ηλεκτρονικής ε, σήμανσης θέτουμε σε κίνδυνο την εκτροφή προβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ε, υπάρχουν οι απαιτήσει για την ηλεκτρονική σήμανση και πρέπει να δούμε ε, αν πρέπει να τις, να διατηρήσουμε ή μήπως μπορούμε να έχουμε ένα πολύ απλούστερο σύστημα. Πάντως, ο χρόνος πιέζει Υπάρχουν ε, ε, πολλά προβλήματα που έχουν ε, δημιουργηθεί. Έχει τεθεί σε ισχύ αυτή η διάταξη και πρέπει οι εκτροφείς προβάτων από την αρχή του έτους να τηρούν αυτές τις διατάξεις για την ηλεκτρονική σήμανση. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν μεταφέρει σε εθνικό δίκαιο αυτή την νομοθεσία είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων, διότι βλέπουν τα τεχνικά ή ε, άλλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν και ακριβώς επειδή υπάρχουν ε, όλες αυτές ε, οι δυσκολίες, ως πολιτική ομάδα προτείναμε να μπει στην ημερήσια διάταξη και να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ ότι είναι δυσανάλογο αυτό το μέτρο, δεν οδηγεί σε αποτελεσματικότητα, είναι πάρα πολύ δαπανηρό και είναι αντιπαραγωγικό και επιζήμιο για την ε, παραγωγή προβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ανιώχη, το λόγο. Thank you, Chairman. Although this regulation... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου ε, τρέχοντος έτους και παρότι ξεκίνησαν αμέσως οι διαμαρτυρίες των ε, παραγωγών, ε, ε, καθυστερήσαμε να συζητήσουμε το θέμα γιατί τα αρνιά τα οποία γεννήθηκαν Ιανουάριο ε, Φεβρουάριο ε, πουλήθηκαν χωρίς ε, να υφίστανται αυτό το σύστημα της ηλεκτρονικής σήμανσης. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πλέον και κάποια στοιχεία μετά το εξάμεινο και δεν είναι απολύτως ικανοποιητικά. Μπορούμε να έχουμε όχι ιδιαίτερα καλή αποτελεσματικότητα. Στην Βρετανία πρέπει να πω ότι έχουμε μεγάλα κοπάδια τα πολυπληθή κοπάδια είναι πολύ ε, συνηθισμένα στην, ε, ε, στη χώρα μου. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία μπορούν να συζητηθούν. Το πρώτο σενάριο βασίζεται μονάχα στον αριθμό των κοπαδιών και βεβαίως θα πρέπει κάποιος να ψάχνει κάθε φορά όλα τα υπόλοιπα αρνιά του κοπαδιού για να δει ε, σε ποιο δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Και μιλάμε για κοπάδια τριών και 4.000 ε, ζώων. Επίσης ε, πρέπει να πούμε ότι στην Βρετανία έχουμε πάρα πολύ μεγάλα, μεγάλες αγορές ζώντων ζώων. Ε, και επομένως εάν ε, η επιτυχία του συστήματος φτάνει στο 96% τότε θα έχουμε πολλά προβλήματα. Δηλαδή θα υπάρχουν ζώα τα οποία θα είναι μη ε, ζώα, δεν θα αναγνωρίζεται η ύπαρξή τους. Το τρίτο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι είναι το 1% της ε, πιθανότητας δειγματοληπτικού ε, διασταυρούμενου ε, ελέγχου. Και θα υπάρξουν σε περίπτωση αποκλήσεων πρόστιμα, δεν το γνωρίζουμε. Ε, βεβαίως δεν είναι απαραίτητο να έχει κανείς την, το ενότιο, μπορεί να έχει ένα άλλο σύστημα σήμανσης. Βεβαίως οι Ισπανοί κέρδισαν χτες ε, στο ποδόσφαιρο, αλλά ε, είχαν ανακαλύψει πριν πάρουν ε, το, το, παγκόσμιο πρωτάθλημα ότι στην κτηνοτροφία εάν πάρεις δώσει επιδοτήσεις στις μικρές μονάδες ή στις μικρές κατσίκες αυτές έχουν κάθε πιθανότητα να πεθάνουν. Απ' την άλλη πλευρά ε, επαναλαμβάνω, εάν το σύστημα επιτυγχάνει μόνο κατά 96%, τι γίνεται με το 4% που δεν καταγράφεται. Ο κύριος Νίκολσον. Ε, θέλω να πω ότι δεν διαφωνώ με αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Απλώς θα ήθελα τα κράτη-μέλη, όταν το συζητούσαμε αυτά τα θέματα τα τελευταία χρόνια, να είχαν καταλάβει τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζαν με αυτό το σύστημα. Θυμάμαι ότι στην Επιτροπή μας κάναμε συζητήσεις και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου και θυμάμαι ότι είχα πει τότε ότι γραφειοκράτες θα το έχουν ε, σχεδιάσει αυτό το σύστημα που ζουν στον πάνω-πάνω όροφο του κτηρίου και δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει το να έχει κανείς ένα κοπάδι με πρόβατα. Δεν μπορεί να το έχει σχεδιάσει αυτό το σύστημα κάποιος που πραγματικά ξέρει τι κάνουν οι παραγωγοί και τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά πέρασαν τώρα απόφαση έχει ληφθεί. Και είπε ο πρόεδρος ότι υπήρχε ένα πρόβλημα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Υπάρχει πρόβλημα διότι η Ιρλανδία δεν έχει εφαρμόσει την ηλεκτρονική σήμανση. Οι δικοί μας αγρότες έχουν εφαρμόσει την ηλεκτρονική σήμανση και τους κοστίζει μία, μία μισή λίρα να να αγοράσουν αυτό την ετικέτα και είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι το σύστημα είναι 96% αποτελεσματικό. Αν, βάλουμε, αν φέρουμε λοιπόν 100, στην, 100 αρνιά στην αγορά, τα 96 θα τα αναγνωρίσουν, τα 4 δεν θα τα αναγνωρίσουν, θα είναι μη αρνιά. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Εγώ συμφωνώ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι έχει ληφθεί η απόφαση μετά από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει και πρέπει να δούμε ε, ε, τι θα κάνουμε όπως ε, συζητάμε και το τι θα κάνουμε με τις κλοποστοιχίε και τους νεοσούς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τι θα κάνουμε τώρα, θα δοθεί παρέκκληση, θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, δεν θα εφαρμοστεί. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι στις περιοχές της δικές μας, στη Σκωτία, στην Ουαλία, όπου υπάρχουν πάρα πολλά πρόβατα και από όπου εξάγουμε πάρα πολλά αρνιά στο εξωτερικό για σφαγή, για να καταναλωθούν σε άλλες χώρες, θα πρέπει να, να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί αν προέρχεται κανείς από κράτος μέλος που δεν εξάγει αρνιά σε άλλη χώρα, λίγο το ενδιαφέρει, δεν του ενδιαφέρει η ηλεκτρονική σήμανση, μπορούν και να μην την χρησιμοποιήσουν. Οι χώρες όμως που έχουν μια προς εξαγωγή ε, ενδιαφέρονται. Γι' αυτό χρειάζεται σαφήνεια σε αυτήν την κατάσταση. Ακόμη και αν 96% αποτελεσματικό το σύστημα, το πρόβλημα είναι ότι οι αγρότε στη δική μου, οι κτηνοτρόφοι στη δική μου χώρα, ταξόδεψαν αυτά τα χρήματα για να προσαρμοστούν με αυτό το σύστημα. μέσα σε μια εβδομάδα χρειάστηκε να αγοράσουν αυτές τις ηλεκτρονικές ετικέτες γιατί ξαφνικά το διαπίστωσαν ότι χρειάζονται αυτές τις ηλεκτρονικές ετικέτες και έτρεξαν να τις αγοράσουν και πάση περιπτώσει ε, τώρα πια ε, το σύστημα το εφαρμόσαμε. Ε, την Επιτροπή την είχαμε ειδοποιήσει ότι δεν είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα, δεν είναι Δεν καταφέρνει κανείς τίποτα παρά μόνο μεγαλύτερη γραφειοκρατία και πλήρη περιφρόνηση από τους γεωργούς για αυτά τα οποία κάνουμε εμεί εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκολσον. Κύριε Μακίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αποσαφημίσουμε ότι δεν υπάρχουν ε, ιδιαίτερα προβλήματα μεταξύ ε, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, κυρίως την 12η Ιουλίου, Τζίνα. Απλώς ε, οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και ισχύουν διαφορετικά προγράμματα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό που σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην ε, Ιρλανδία, ε, είναι ότι γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί η κοινωνική εξαίρεση. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα ζώα μέχρι 12 μηνών εξαιρούνται από αυτήν την ηλεκτρονική σήμανση και ενδεχομένως και ορθώς η Ιρλανδική εκδοχή και εξήγηση είναι πιο σωστή και πιο καλή ε, φιλική για τον ε, χρήστη. Όμως ελοχεύει ένας κίνδυνος. Προχωρώντας, πρέπει κάποια στιγμή κάποια πράγματα να εφαρμοστούν ταυτόχρονα από όλους και ο κύριος ε, Νίκολσον αναφέρθηκε και στο θέμα της ευζοίας των ζώων. Κοιτάξτε, εάν δεν εφαρμόσουν όλοι ταυτόχρονα ε, την ίδια νομοθεσία, τότε πράγματι φτάνουμε σε αδικίες. Κάποιοι έχουν ήδη πάρει χρήματα και τα έχουν χρησιμοποιήσει για να εφαρμόσουν αυτούς τους ε, κανόνες. Ε, εν πάση εγώ δεν βλέπω να αλλάζει η άποψη για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το σύστημα να αποβεί λειτουργικό και σωστό ε, και τελικά θετικό για τους κτηνοτρόφους με την έννοια ότι θα αποφευθούν αρρώστιες κτλ. Θα ήθελα πάντως να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά ε, την πολλαπλή συμμόρφωση ε, για το σύστημα αυτό. Γιατί διαφορετικά όντως θα δημιουργηθούν προβλήματα σε ορισμένους κτηνοτρόφους σε διαφορετική περίπτωση. Ο κύριος Λάιον. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι και άκουσα από τον κύριο Γιάρ ε, ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη, γιατί άρχισα να πιστεύω ότι μόνο η αντιπροσωπή του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ανησυχούσε τόσο πολύ για αυτό το θέμα. Ήταν ε, μια αντίδραση την οποία είχαμε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο για ε, ε, ε, το μέτρο αυτό και ο συνάδελφος είπε ότι το είχατε συζητήσει και σε προηγούμενες θητείες του Κοινοβουλίου, πολύ πριν έρθω εγώ στο Κοινοβούλιο. Πάντως εδώ η τεχνολογία δεν μπορεί να μας δώσει 100% αξιοπιστία του συστήματος Μιλάνε για 92-94% αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε το, το, το 100% για τις αγορές, για τα παζάρια των ζώων, των ζώων. Όταν φτάνουν 7.000 ε, και έχουμε ένα 10% σφάλμα, θα υπάρχουν ε, το 10% των ζώων που δεν θα έχουν καταγραφεί τι κάνουμε και σε περίπτωση που έχουμε κρούσμα κάποιας ζωονόσου, πώς θα κάνουμε την ανείχνευση των ζώων τα οποία πουλήθηκαν. Η τεχνολογία δεν μπορεί να μας δώσει ακρίβεια 100%. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τον κλάδο έναντι πιθανού κρούσματος ζωονόσου για να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε το ζώο από το οποίο ξεκίνησε ε, κάποια νόσος. οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι είναι στο έλεος της τεχνολογίας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πολλαπλή συμμόρφωση και αν φτάσουν το 90% στην συμμόρφωση φταίνε αφού θα, έχει, θα έχουν υποστεί τις συνέπειες ενός συστήματος το οποίο λόγω της τεχνολογίας δεν μπορεί να, να, να τους καλύψει 100%. Πιστεύω ότι είναι άδικο λοιπόν αυτό για τους κτηνοτρόφους και πρέπει να το αναγνωρίσει η Επιτροπή και τουλάχιστον να συμφωνήσει για κάποια αμνηστία τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του συστήματος με σκοπό να επανεξετάσει την πρακτική εφαρμογή του συστήματος, να εξετάσει τον κανονισμό και αντί να κάνει αυτό που έκανε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και να λέει αυτό θα γίνει και τελεία, να δείξει κάποια προθυμία να ακούσει τα ειλικρινή παράπονα των κτηνοτρόφων, γιατί είναι η πραγματικότητα ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να καλύψει αυτούς τους κτηνοτρόφους. Θέλουμε λοιπόν μια υπόσχεση από την Επιτροπή ότι θα επανεξετάσουν αυτό το θέμα και θα κάνουν ένα ειλικρινή διάλογο με τον κλάδο των κτηνοτρόφων για το τι μπορεί να γίνει. Ε, να μην απαντήσει η Επιτροπή αυτό που απάντησε στους συναδέλφους των ε, κ. Νίκολσον και τον άλλο συναδέλφο που μίλησε ότι αυτό πρέπει να γίνει και τελεία. Περιμένουμε από την Επιτροπή κάποια κατανόηση. Ο κ. Άλαν Σμιτ Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγα είναι τα θέματα στα οποία όλες οι νήσοι του αρχιπελάγους ε, είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Ε, συγχαρητήρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τελικά καταφέρατε οι Σκοτσέζοι, οι Ουαλοί, οι Άγγλοι να έχουν ε, κοινή αντίδραση. Ήδη από την προηγούμενη θητεία είχαμε πει ότι χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στην Επιτροπή και χωρίς να θέλουμε να κάνουμε έτσι κακό διάλογο, ε, είχαμε προειδοποιήσει, λέω, ότι δεν θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Ε, το σύστημα πρέπει να είναι πάντα λογικό και πρέπει να είναι πάντα ε, λογικό. Επίσης, ε, μας ε, έλεγαν ότι στο Συμβούλιο μόνο εμείς δεν είχαμε συμφωνήσει μέχρι τώρα, όλοι οι άλλοι το έχουν κάνει, αλλά αυτά είναι φαντασιώσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στις άλλες ε, χώρες που το έχουν εφαρμόσει. Υπάρχουν δε πάρα πολλέ χώρες οι οποίες δεν έχουν καν εφαρμόσει το σύστημα αυτό, έχουν ζητήσει εξαιρέσεις κτλ. Στην Σκοτία χάσαμε βεβαίως τη συζήτηση, αλλά παρόλα αυτά γίνεται μια προσπάθεια η Σκοτία προσπάθησε να εφαρμόσει τον ε, κανονισμό αυτό. Και τελικά το, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε φτάσει είναι το 93%. Ε, αυτό σαν αποτέλεσμα ορθότητας βεβαίως είναι εξαιρετικά υλικές και παραμένει ένα 7% το οποίο ε, τι γίνεται. Ε, ναι, βεβαίω, όλοι γνωρίζαμε και εκ των προτέρων ότι υπάρχουν προβλήματα ε, τεχνικά και η Κομισιόν το ήξερε. Καταλαβαίνετε τον ε, προβληματισμό μας και, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να δούμε και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά την επιβολή ε, των ε, κανόνων. Ε, τι να σας πω, εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι θέλουν να εγκαταλείψουν το, τον χώρο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι απογοητεύονται από την κατάσταση. Και βεβαίως αυτό αποτελεί και πλήγμα κατά την άποψή μου ε, ένα πλήγμα ε, για την συνολική αντιμετώπιση της κοινής γεωργικής πολιτικής και χαίρομαι που ο συνάδελφος ε, έφερε το θέμα αυτό. Δηλαδή πιστεύουμε ότι τελικά αμαυρώνεται ολόκληρη η κοινή γεωργική πολιτική. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν πρόκειται να βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει πιο ελκυστική. Είναι ένα αντιευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα εντείνει τον ευρωσκεπτικισμό. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν καλύπτει τον σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί, καλύτερα να μην το εφαρμόσουμε μέχρι τη στιγμή που θα μπορούμε να το κάνουμε, να το εφαρμόσουμε σωστά. Ε, είναι καλό που η συζήτηση αυτή γίνεται σήμερα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναληφθεί η συζήτηση αυτή και στο μέλλον στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να λάβω το λόγο, αλλά μόνο με χιούμορ μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα της ηλεκτρονικής ε, σήμανσης. Ε, αυτά τα ποσοστά που αναφέρθηκαν, ότι το 96% μπορεί να είναι αποτελεσματικό και το 4% ε, να μην είναι, τι το κάνουμε αυτό το 4%? το ίδιο ισχύει και με συστήματα ε, για τα βοηδή. Κάποιος είχε μια γελάδα, μια μόνο γελάδα που κούσε κάπου στα βουνά. Είχε μία και μόνο γελά. Δεν είχε ακούσει ποτέ για ε, σύστημα ε, ηλεκτρονικής σήμανσης και δεν ε, και δεν ε, μπορούσε να την πουλήσει γιατί δεν, ήταν, δεν είχε το σύστημα της ηλεκτρονικής σήμανσης. Ε, δεν μπορούσε να την κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να την πουλήσει επειδή δεν είχε το σύστημα της ηλεκτρονικής σήμανσης ε, και την πήγε στον κτηνίατρο ε, ε με σκοπό να την κοιμήσουν γιατί ισχυρίστηκε ότι είχε σπάσει το πόδι της η Αγελάδα και έπρεπε να την ε, κοιμήσει ε, ε, θανατώσει επομένω ο, ο κτηνίατρος. Και δεν μπορούσαν να βρουν μια λύση για το τι θα κάνουν ώστε να μπορέσει να πουλήσει, να, να βγάλει κάποια άκρη με αυτή τη μία και μόνη αγελάδα που είχε αυτός ο κτηνίατρος. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή. Όταν φτάνουν αρνιά από την Αυστραλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 100% εγγυημένη η χνηλασιμότητα του πρόβιου κρέατος από την Αυστραλία, ώστε να ζητάμε 100% από την, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 6.30 πρέπει να εγκαταλείψουμε την αίθουσα. Θα δώσουμε τον λόγο στην ε, Επιτροπή και μετά έχουμε και συνάντηση των ε, συντονιστών. Άρκιν, Ρόντουστ και μετά Επιτροπή. Πολύ σύντομη. Γιατί νομίζω ότι όλα ε, τα είπε κανεί, τα, όλα υπόθηκαν. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι σαφές. Δεν έχει δώσει η τεχνολογία ε, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα της του 95-96%. Παραμένει ένα 5-4% τι θα γίνει με αυτά τα ζώα. Πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν λειτουργεί καλά το σύστημα αυτό. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχει μία ε, μία ε, εξαίρεση στην Ιρλανδία για όσον αφορά τα σφαγεία ε, για τα ε, ζώα μέχρι 12 μηνών. Ε, και, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε μονάχα για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία. 14 ε, εκατομμύρια ζώα αρνιά έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία και επομένως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με αυτά τα ζώα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πολύ βέβαιη ότι το σύστημα λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πολύ για όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ και έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε ήδη πόσοι κτηνοτρόφοι έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητα και έχουν ε, σταματήσει ε, να εκτρέφουν τα κοπάδια τους. το Σλέσφιχ και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι σημαίνει για τον ε, κλάδο και τι σημαίνει για τις δραστηριότητες σε όλες τις περιοχές. E Ευχαριστώ κύριε Ρόντουστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ο δόκτωρο Ντομάδα. Θα πρέπει να κάνω μία ιστορική αναδρομή για αυτό το θέμα το οποίο δημιουργεί μεγάλη δυσαρέσκεια. Πρώτον, η απόφαση αυτής ε, της, ε, για την εισαγωγή ε, της ηλεκτρονικής σήμανσης, μονομένου συστήματος δηλαδή η ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων, ελήφθη από το Κοινοβούλιο, με σύμφωνο γνώμη του Κοινοβουλίου το 2003, μετά από την κρίση του αυθόδους πυρετού. Τότε ο κανονισμός 21 του 2004, του Ιανουαρίου δηλαδή του 2004, προέβλεπε ότι η μεμονωμένη ε, ίχνη λασιμότητα και η μεμονωμένη ατομική ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων, των εγωπροβάτων, θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Όμως, θα μπορούσε να υπάρξει ε, πιθανή τροποποίηση μετά από έκθεση και εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή ενέκρινε την ε, πρόταση και την ε, έκθεση, δεν ε, ανέφερε καμία συγκεκριμένη ημερομηνία όσον αφορά το σύστημα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής σήμανση των προβάτων. Όμως, αντιθέτω, πρότεινε να αποφασιστεί η ημερομηνία μέσα από διαδικασίες επιτροπολογίας μετά από την γενικότερη αξιολόγηση και μελέτη επιπτώσεων η πρόταση της Επιτροπής δεν έγινε δεκτή από το Κοινοβούλιο, ούτε όμως και από το Συμβούλιο, το οποίο το, 2007, το 2007, ευθυγραμμιζόμενο με την θέση του Κοινοβουλίου, όρισε ε, σαν ημερομηνία εισαγωγής του συστήματος ηλεκτρονικής ε, υποχρεωτικής ε, σήμανσης των προβάτων την 1η Ιανουαρίου του 2010. Τι ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευθυγραμμιζόμενη με την πρόταση του Κοινοβουλίου. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισε ε, μέσω της μέγιστης χρήσης ε, της ευελιξίας ε, του ιδίου κανονισμού διασφάλισε, λέγω, ένα μεγάλο αριθμό εφαρμοστικών κανόνων έτσι ώστε βαθμιαία να αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα και επίσης ε, εισήγαγε και περαιτέρω ευελιξία, ας πούμε επιτρέποντας ότι η ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων ε, να γίνεται ας πούμε ε, στην, στο τελικό προορισμό των ζώων ας πούμε στην αγορά ή στο σφαγείο και όχι στην εκτινοτροφική μονάδα. Όμως, όπως γνωρίζετε από την 17η Ιανουαρίου υπάρχει μια σειρά υποχρεωτικών μέτρων σε πολλές ε, χώρες. Κατά αυτή την έννοια πρέπει να πω ότι ο κανονισμός προέβλεπε ότι τα κράτη-μέλη, εάν το επιθυμούσαν, θα είχαν την δυνατότητα να εισάγουν βαθμαία το σύστημα ε, ήδη πριν από το 2010. Επομένως, και σε σχέση με τα προβλήματα ανάμεσα στην ε, Δημοκρατία της Ιρλανδίας ε, και την ε, Βόρεια Ιρλανδία μπορούσαν να προβλεφθούν διαδικασίες έγκρισης οι οποίες ενδεχομένως οδηγούσαν σε κάποια προβλήματα λόγω πρώιμης εφαρμογής. Όμως, το γεγονός ότι ο κανονισμός αυτός αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης αντιπαράθεσης, δεν οδήγησε ε, στην σωστή βαθμία εφαρμογή του και εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα ε, για τις ε, χώρες αυτές ε, οι οποίες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν ως μέχρι τελευταία στιγμή τις προθεσμίες που προέβλεπε ο κανονισμός. Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα έχουν λυθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 που είναι η τελική ημερομηνία έγκρισης των μέτρων αυτή τη, σε αυτή την ημερομηνία οι κτηνοτρόφοι θα έχουν την υποχρέωση ε, για πλήρη ηλεκτρονική σήμαση των προβάτων, αλλά όχι και για την πλήρη ηχνηλασιμότητα. Βεβαίως, ε, εμείς ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι όλα τα τεχνικά προβλήματα τα οποία διαφάνησαν τα τελευταίους μήνες θα λυθούν. Βεβαίως, δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι εάν εάν το σύστημα λειτουργήσει μονάχα ε, στο 96%. Πρέπει να πω πάντως ότι η ηλεκτρονική σήμανση των ε, ζώων λειτουργεί ταυτόχρονα με τα παραδοσιακά ενότια. Και σε περίπτωση που το σύστημα το ηλεκτρονικό δεν λειτουργήσει υπάρχει ε, το άλλο σύστημα. Βεβαίως είναι γεγονός ότι όταν το ποσοστό λάθους ή αποτυχίας είναι ψηλό, τότε ε, αποτυγχάνει και η ευκολία που συνεπάγεται το ηλεκτρονικό σύστημα και με την ε, μεμονωμένη ε, εναλλακτική λύση του παραδοσιακού συστήματος χάνονται όλα τα προτερήματα του ηλεκτρονικού συστήματος. Πάντως θεωρούμε ότι υπάρχουν όλα τα εχέγγυα ε, ώστε το σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα να εφαρμοστεί σωστά και ε, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες αποστολές επιτόπου ε, ανιχνευτικές, τις οποίες ονομάζουμε fact-finding missions, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Το, ζήτημα της συχνηλασιμότητας πρέπει να πω ότι έχει λυθεί. Δηλαδή ε, υπάρχει ένα ισχύον σύστημα, ιδιαίτερα δαπανηρό, ε, χάρτινων διαβατηρίων ε, τα οποία διασφαλίζουν την απόλυτη χνηλασιμότητα όσον αφορά τα βόια, ε, το βόλιο κρέας. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για την πολλαπλή συμμόρφωση. Διαβάζω μία φράση από τα έγγραφα, και της, από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το σύστημα ενωτίων των ε, βοήων. Ένα έγγραφο το οποίο βοηθάει τους ελεγκτές, τους επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ελέγχουν την πολλαπλή συμμόρφωση. Αναφέρομαι στην, ε, στα ενότια, τα παραδοσιακά ενότια και διαβάζω στα αγγλικά. δυσκολίες, ε, ε, προβλήματα ε, μπορούν να υπάρξουν και εάν δεν ξεπερνούν ένα λογικό περιθώριο λάθους δεν θα υποβάλλονται, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και στο παραδοσιακό σύστημα προβλέπονται κάποια περιθώρια λάθους και οι υποδείξεις που γίνονται, οι οδηγίες που δίνονται στους επιθεωρητές είναι ότι όταν το λάθος αυτό αποτελεί ένα λάθος τεχνολογίας, ένα λάθος ε, απλό από αυτά που μπορούν να συμβούν ε, μετά από μεγάλο ρυθμό συναλλαγών, τότε το λάθος αυτό δεν θα προκαλεί κυρώσεις. Βεβαίως στο μέλλον θα συζητήσουμε και με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας όλα τα θέματα αυτά ε, και ε, όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα πολλαπλής συμμόρφωσης και να δούμε εάν τα συστήματα πολλαπλής συμμόρφωσης για το τομέα του βοήου κρέατος μπορεί να εφαρμοστεί ε, στο, στο τομέα των εγωπροβάτων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τώρα τις εργασίες της Επιτροπής μας. Είναι η τελευταία μας συνάντηση, ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν θα είσαστε όλοι εδώ 19 και 20 Ιουλίου. Α, έχουμε αύριο το πρωί, έχετε δίκιο, λέει ο πρόεδρος. Ναι, ξεχάστηκα, ξεχάστηκα. Αύριο το πρωί, λοιπόν, θα ξανασυναντηθούμε. Αύριο το πρωί θα ακούσουμε βεβαίως και τον εκπρόσωπο της Βελγικής Προεδρίας. Ζητώ συγγνώμη. Ε, τώρα όμως θα συνεδριάσουν οι